Good morning, colleagues. It's o'clock. Καλημέρα σας. Είναι νέα, οπότε μπορούμε να αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Καλώς ήρθατε. Και καλώς ήρθαν ε, και όσοι παρακολουθούν από το διαδίκτυο την συνεδρίασή μας. Καλώς ήρθατε όπου και αν βρίσκεστε στην ε, Ευρώπη. Έχουμε πολλά θέματα για σήμερα, οπότε θα δουλέψουμε μέχρι σήμερα το απόγευμα, μην καθυστερήσουμε άλλο, συνεπώς. Για τη συνεδρίαση των συντονιστών τώρα, θα ήθελα να σας πω που καταλήξαμε. Και συγγνώμη αν δεν είναι πολύ ενδιαφέροντος, θα σας πω και θα διαβάσω διάφορα νούμερα, αλλά έτσι πρέπει να κάνω. Λοιπόν, εγκρίθηκε η ημερήσια διάταξη για το Σεπτέμβριο. Αυτό ήταν το πρώτο θέμα. Εγκρίθηκε λοιπόν η μερίσια διάταξη για την 7η Σεπτεμβρίου που συμπεριλαμβάνει τις 0099, 01038, 141 0141, 0151 και 155. 13.04, μηδέν 048 και 1525 θα μπουν στην εμερήσια διάταξη του Οκτωβρίου. Όλα, αυτά τα θέματα βέβαια θα μπουν στην ημερήσια διάταξη εφόσον έχουμε τις απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν δεν έχουμε έγκαιρα απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναβληθούν. Για τις συστάσεις για τις οποίες υπήρχε ένσταση. Η 0163 και 0176 εγκρίθηκε η δικιά μου σύσταση και έκλεισαν οι αναφορές αυτές. 0148 του 2017 παραμένει ανοιχτή και θα στραφούμε στην Επιτροπή για πρόσθετες πληροφορίες και όλες οι άλλες εγκρίθηκαν σύμφωνα με τους συμβασμούς που πρότεινα εγώ. Για τα θέματα Β, θα δείτε όλες τις αποφάσεις που συμπεριλαμβάνουν το, στα πρακτικά. Τώρα για τις ερευνητικές μας ε, επισκέψεις. Είπαμε, Τάραντ, την επόμενη εβδομάδα και το Σεπτέμβριο στη Λάρνακα. Ακρόαση για την προστασία των προσωρινών εργαζομένων και των δικαιωμάτων τους θα μεταβληθεί ο τίτλος ω εξής. Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων οι οποίοι απασχολούνται σε προσωρινή απασχόληση σε επισφαλή απασχόληση. Οι συντονιστές ε, ε, κλήθηκαν επίσης να προτείνουν για το πρώτο εξάμενο του 2018 ε, επισκέψεις ερευνητικές και αυτό έχουν να το κάνουν μέχρι το Σεπτέμβριο. Για το Brexit θα παρακολουθήσουμε όλες τις αναφορές οι οποίες έχουν βρεθεί στην ημερήσια διάταξη της 21ης Ιουνίου για παράδειγμα όλες που έχουν να κάνουν με το Brexit λοιπόν. Και όπως ζήτησε μία ομάδα θα ζητήσουμε ένα ψήφισμα, ένα σύντομο ψήφισμα για αυτό το θέμα. Η Γκουέ ζήτησε να εκπονήσουμε και έκθεση για τις υποθήκες και για την στέγαση βάσει των αναφορών που έχουμε λάβει μέχρι τώρα. Και είπαμε ότι θα υποβάλουμε ε, ερώτηση προφορική στην Κομισιόν χωρίς ψήφισμα για να δώσουμε συνέχεια στο ψήφισμα το οποίο ανέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2015 για το ίδιο θέμα. Οι συντονιστές επίσης αποφάθηκαν υπέρ του να στραφούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ενημερώσει για μελέτη που ετοιμάστηκε από τη ΛΥΜΠΕ το 2015 για την οδηγία όσον αφορά την υποβοήθηση θα υπάρξει κάποια συνέχεια λοιπόν θα δώσουμε και θα έχουμε και μεικτή συνάντηση με την Επιτροπή Γυναικών, κυρίως για το θέμα της βίας σε βάρος των γυναικών. Συμφωνήσαμε οι συντονιστές να ψάξουμε να βρούμε και άλλους τρόπους για να συνεργαστούμε καλύτερα και πιο πολύ με την Επιτροπή Γυναικών και θα οργανώσουμε κοινέ συνεδριάσεις για θέματα που απασχολούν και τις δύο επιτροπές όπως ήταν αυτό. Επίσης ενημέρωσα προφορικά για το τι γίνεται στην Επιτροπή Προέδρων ε, Επιτροπών, όπου προεδρεύω εγώ. Εκεί έχουμε συζητήσει για τη δήλωση της Ρώμης, για τη διοργανική συμφωνία για την καλύτερη νομοθέτηση και τέλος για την αναθεώρηση του εγχειριδίου όσον αφορά την αξιολόγηση αντικτύπου. Επίσης, οι συντονιστές σημείωσαν ότι υπήρξε ε, συνεδρίαση σε επίπεδο προσωπικού του δικτύου αναφορών στις 16 Ιουνίου και αντίστοιχη συνάντηση θα υπάρξει σε επίπεδο Ευρωβουλευτών στις 10 ε, Οκτωβρίου. Αυτά περί συντονιστών χτες. Οπότε, περάσουμε στο σημείο 13 στην ημερήσια διάταξη Πρόκειται για την αναφορά 178. Πρόκειται για την εφαρμογή συνθηκών απασχόλησης και προπτικών σταδιοδρομίας που δεν εισάγουν διακρίσεις για τους έκτακτους και τους συμβασιούχους ή υπαλλήλους στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Πρώτα απ' όλα καλωσορίζω εδώ τον κύριο Μάικλ Άσπρουκ που είναι αναφέρον. Και θα σας δώσω το λόγο για πέντε λεπτά παρακαλώ. Good morning. Um, I hope... Καλημέρα σας. Δεν φαίνεται με το τηλεχειριστήριο να μπορώ να μετακινηθώ μέσα στις διαφάνειες, μήπως κάνω κάτι λάθος. Oh, please. I'll have to go up front. Okay. Θα χρειαστεί να πάω μπροστά, ζητώ συγγνώμη. Where do I point it? Προς τα πού πρέπει να είναι στραμμένο, γιατί δεν δουλεύει. Comme ça? Ah, okay, we'll do it with my finger. My finger works a lot better. Με το δάχτυλο καλύτερα. Από ό,τι φαίνεται καλημέρα κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, ε, εκπρόσωποι των ε, ΜΜΕ, πολίτες και οι φίλοι μου που πάσχουν από βεβαιότητα που κάθονται εκεί πίσω. Δεν είμαι εδώ για να γκρινιάξω κατά της Κομισιόν και να πω ότι όλα είναι φρικτά και όλα αυτά. Αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να βελτιώσουμε λίγο παραπάνω τις συνθήκες εργασίας. Να σας αναφέρω συντομία την απάντηση της Επιτροπής στην οποία έχω ήδη απαντήσει και το στείλα και σας ε, την απάντηση με email. Ουσιαστικά Οι απαντήσεις τους καταδάζονται σε δύο κατηγορίες. Από τη μία λένε, κοιτάξτε, το 2013 ο νομοθέτης αποφάσισε το κετό. Αν και αυτή δεν είναι πλήρης απάντηση, πρέπει να μας εξηγήσουν γιατί δεν μπορούμε να το βελτιώσουμε αυτό το 2017. Και ξέρετε, έχουν γίνει πολλά, έχουν παρευληθεί πολλά μετά του, μεταξύ του 2013 και του 2017, έτσι δεν είναι. Κάτι άλλο είναι ότι απορρίπτουν πράγματα τα οποία εμείς δεν ισχυριζόμαστε καν. το να πετάμε με ανθρώπους έξω μετά από έξι χρόνια πρακτικής εμπειρίας είναι μια τεράστια σπατάλη πόρων. Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί το ακριβές ποσό, αλλά μιλάμε πιθανότητα για χιλιάδες ευρώ για κάθε ε, προσωρινά εργαζόμενο, για κάθε έκτακτο εργαζόμενο. Θα ήθελα να επισημάνω εδώ ότι και αντίθετα από κάποια πράγματα που θεωρούνται δεδομένα, ε, ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων εφαρμόζεται και σε εμάς ε, που εργαζόμαστε στα θεσμικά όργανα. Αυτό φαίνεται σαφώς στην απόφαση του δικαστηρίου, ε, στην απόφαση Στρακ και η Κομισιόν έχει μαχηθεί κατά αυτής της απόφασης αυτής που λέει ότι κάποιοι άνθρωποι μπορούν να επικαλεστούν το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και όπως βλέπετε έχουν χάσει άσχημα έχουν φάει ξύλο από το δικαστήριο, για να το πω έτσι. Και το δικαστήριο του είπε πρέπει να πληρώσετε και τι δικέ σα δαπάνε και των αλλανών. Μιλάμε για μεγάλο χαστούκι. Οπότε ήταν πολύ σαφή η απόφαση του δικαστηρίου. Κάτι άλλο που πρέπει να σας πω νομικά είναι η οδηγία για την εργασία ορισμένου χρόνου. Ε, που απευθύνεται στα κράτη-μέλη και η Κομισιόν λέει ότι εμείς δεν είμαστε κρατός μέλος, αλλά πώς εξηγείτε ότι ισχύει για όλους πέραν αυτού που συνέταξε την οδηγία που συμμετείχε στη δημιουργία της και πώς μπορείτε να εξηγήσετε ότι αυτές οι αρχές της οδηγίας δεν ισχύουν για τους δικούς τους εργαζομένους. Δεν νομίζω ότι μπορείτε να ισχυριστείτε κάτι τέτοιο, ούτε να το εξηγήσετε. Και πιστεύω ότι αυτή η οδηγία για την εργασία ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με αυτήν ε, οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου έχουν όλα τα ίδια, ε, έχουν τα ίδια ε, πλεονεκτήματα με αυτούς τους όρους του χρόνου, εκτός από τα προράτα. Οπότε και οι εργαζομένοι ορισμένου χρόνου θα πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες να μονιμοποιηθούν. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται διακριτική μεταχείριση το οποίο είναι το αντίθετο από αυτό που λέει η Κομισιόν. Η Κομισιόν λέει ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να του δίνουμε τα ίδια δικαιώματα σε κανένα τομέα. Πάντα πρέπει να του έχουμε λίγο χαμηλότερα. Πρέπει να διατηρούμε το σύστημα με τι κάστε. Και εγώ θέλω να κάνω μία ε, συναισθηματική εδώ έκκληση για να καταλάβετε τι σημαίνει να δουλεύει κανείς με σύμβαση ορισμένου χρόνου και να ξέρετε ότι ε, τρέχει αντίστροφη μέτρηση και ξέρει ακριβώ τη χρονική στιγμή που θα βρεθεί χωρί δουλειά και δεν έχει σημασία. Μπορεί να πάρει ε, και βραβείο Νόμπελ. Και σε αυτή την περίπτωση ακόμη θα σε πετάξουν έξω. Το δεύτερο σημαντικό κομμάτι τη ε, αναφορά στο πρώτο είναι να σταματήσουμε αυτέ τι ανοησίε του να απολύουμε κόσμο μετά από 6 χρόνια, ακόμη και αν οι επιδόσει του ήταν άρεστε. Μερικέ φορέ και καλύτερε από τον μονίμων. Το άλλο που θα θέλαμε ας ανοίξουμε τους εσωτερικούς διαγωνισμούς στους ε, συμβασίους ορισμένου χρόνου. Έχουμε κάνει κάποια βήματα στην Επιτροπή σας με την αναφορά την 192. Ελάχιστοι θα με θυμάστε από τότε, αλλά η Κομισιόν εξακολουθεί να μας κρατά σε απόσταση. Πρέπει να βιαστώ τώρα, λέτε, να επιταχύνω. Αυτό είναι σημαντικό, διότι οι εσωτερικοί διαγωνισμοί έχουν προς το επιτυχίες 25% Οπότε ένα πολύ σημαντικό δικαίωμα το να μπορεί κανείς να συμμετέχει σε τέτοιους διαγωνισμούς. Και μετά ξέρετε όλη τι σημαίνει επισφαλής εργασία, αβέβαιη εργασία. Ξέρετε πόσο βλάπτει την Ευρώπη, δεν χρειάζεται να το επαναλάβω. Σε τελική ανάλυση το μόνο που ζητάμε είναι λίγη παραπάνω δικαιοσύνη. Δεν ζητάμε απόλυτη δικαιοσύνη. Εδώ βλέπετε τα στοιχεία μου. Σας ευχαριστώ. And we thank you very much. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Σας διαβεβαιώ δεν συμβαίνει συχνά να χειροκροτάει το κοινό κάποιον αναφέροντα. Είναι κάτι ασυνήθιστο στην Επιτροπή μας. Τώρα να στραφώ στην Κομισιόν. Έχω πολλά ονόματα. Εσείς θα αποφασίσετε ποιος θα μιλήσει πρώτος. Και αν θέλετε να μιλήσει ένας ή δύο συνάδελφοι από την Επιτροπή, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, κύριε Ασμπρόκ, σας ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία. Ονομάζομαι Ρομπέρτο Καρλίνη και είμαι τμήματάρχης του τμήματος προσλήψεων της Κομισιόν. Δίπλα μου ο κύριος Ροκ, τμήματάρχης ε, του τμήματος νομικών υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπινών Πόρων. Πράγματι Εγώ είμαι ο πρώτος ενδιαφερόμενος ε, όσον αφορά την πρόσληψη συμβασιούχων. Εγώ υπογράφω τις συμβάσεις τους. Ανέκαθεν ε, προσέχαμε ιδιαίτερα τα προβλήματα που ανέφερε ο κύριος Άσμπροκ και προσπαθούμε στο βαθμό του δυνατού να ανταποκριθούμε στις απαιτήσει και των συμβασιούχων ε, προς όφελος φυσικά της υπηρεσίας. Ποιο είναι το όφελος της υπηρεσίας ή συμβασιούχοι ε, εισήχθησαν ως θεσμός το 2004 έχουν περάσει σχεδόν δηλαδή 15 χρόνια από την πρώτη τους εισαγωγή ωστόσο οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου γίνονταν και πριν το 2004 με την ονομασία βοηθητική υπάλληλη ε, πριν το 2004 ανανεώνονταν κάθε μήνα δηλαδή ήταν απόλυτη αβεβαιότητα και η αστάθεια τόσο για την υπηρεσία όσο και για τους εργαζομένους από το 2004 και μετά έγιναν κάποια σημαντικά βήματα προς τα μπρος και το 2014 με την τελευταία ενημέρωση η μέγιστη διάρκεια διπλασιάστηκε από τα 3 στα 6 χρόνια για την απασχόλησή του αυτό για να δοθεί κάποια σταθερότητα τόσο στην υπηρεσία όσο και ε, στον ενδιαφερόμενο, στον ε, εργαζόμενο. Από τη στιγμή φυσικά που έπαιρνε κάποιος, ε, λάμβανε μια σύμβαση, γνώριζε το χρόνο εργασίας του χωρίς αυτό να υποχρεώνει το θεσμικό όργανο να κρατήσει τη σύμβαση μόνο για 6 χρόνια. Ήξερε όμως ο εργαζόμενος ότι στα 6 χρόνια ολοκληρωνόταν η σύμβαση. Αυτό ήταν απόλυτα διαφανές και βέβαιο. Ε, χρησιμοποιούμε συμβασιούχους ορισμένου χρόνου για να καλύψουμε κάποιες ανάγκες ε, υπό δύο έννοιες. Το να δίνουμε μια σταθερότητα στην υπηρεσία αλλά και το να δίνουμε τη δυνατότητα ανανέωσης ε, ε φρεσκαρίσματος κατά κάποιο τρόπο των ε, δεξιοτήτων. Ειδικότερα σε ορισμένους τομείς ε, πιο ειδικευμένους. Για παράδειγμα, Μπορούμε να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις που όλοι γνωρίζουμε στον οικονομικό τομέα, στον τομέα των μεταναστών και σε άλλους τομείς ε, ε, που χαρακτηρίζουν τη σημερινή κρίση. Η ανάγκη αυτή λοιπόν ε, υπήρχε, υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει στο μέλλον. Όσον αφορά τις νομικές πτυχές, χωρίς να θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, ενδεχομένως αυτές θα μπορείς να τις αναλύσει καλύτερο ο συνάδελφός μου, ο κ. Ροκ, ε, θα ήθελα να υπενθυμίσω ε, παραδείγματι ότι χρησιμοποιούμε συμβασίου ορισμένου χρόνου ε, και η κατάσταση αυτή πολλές φορές έχει αποτελέσει το αντικείμενο προσφυγής στο δικαστήριο. Η τελευταία αρκετά σημαντική περίπτωση, αλλά όχι σημαντικότερη που ήθελα να αναφέρω, ήταν η υπόθεση C16 του 2015 της κυρίας Μαρία Λένα Τέρες Λόπες ε, όπου το δικαστήριο υπενθυμίζει ότι όχι μόνο είναι δυνατόν ε, στο, στους δημοσίους φορείς να υπάρχουν συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου, ε, αλλά πρέπει αυτοί να διατηρούνται σε κάποιο πλαίσιο νομιμότητας και ε, γενικότερης ορθότητας. Και στο πλαίσιο αυτό εμείς ε, δείχνουμε σεβασμό τόσο στην διαφάνεια ε, από την πράξη πρόσληψης μέχρι τις ανανεώσεις των συμβάσεων αλλά και στο γενικότερο πλαίσιο διότι ξέρετε η Κομισιόν έχει γενικούς κανόνες μέγιστης παρουσίας των συμβασιούχων της ε, οπότε έτσι θέλουμε να αποφύγουμε άνθρωποι που μπαίνουν ε, με συμβάσει ορισμένου χρόνου και το γνωρίζουν να παραμένουν για υπερβολικά μεγάλο διάστημα και να παραμένουν απομακρυσμένοι από την εξωτερική αγορά, στην οποία θα πρέπει να παραταχθούν για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Το δεύτερο στοιχείο είναι η πρόσβαση ε, στου εσωτερικού διαγωνισμού. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να διευκρινίσω κάποια νούμερα που δεν συμφωνούν ε, με την πραγματικότητα. Όσον αφορά τον αριθμό πτυχιούχων και το ποσοστό επιτυχία στου εσωτερικού διαγωνισμού, για παράδειγμα, στον τελευταίο εσωτερικό διαγωνισμό που έλαβε χώρα, ε, υπήρξαν 3.000 ε, ε, υποψήφοι, 80 ήταν οι τυχιούχοι, πάνω από το, κάτω δηλαδή από το 20% που ανέφερε και ο Σάσμπροκ. Ο νομοθέτης του 2014 έδωσε τη δυνατότητα κατ' εξαίρεση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 82.7, να δίνεται δυνατότητα πρόσβασης ε, των συμβασιούχων σε εσωτερικούς διαγωνισμούς. Ε, το έχουμε κάνει, θα το επαναλάβουμε. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι αυτοί οι εσωτερικοί διαγωνισμοί να έχουν ποσοστό επιτυχία συγκρίσιμο ουσιαστικά με αυτό των εξωτερικών διαγωνισμών που παραμένει το κύριο τρόπος, η κύρια μέθοδος που χρησιμοποιούμε και που θέλουμε να χρησιμοποιούμε για τις προσλήψεις τώρα και στο μέλλον των μονίμων υπαλλήλων. Σας ευχαριστώ και αν υπάρχουν ε, άλλες ερωτήσεις για το νομικό κομμάτι, ο κύριος Ρόκ είναι στη διάθεσή σας. Please go ahead with the legal aspects. Παρακαλώ, μπορείτε να περάσετε στις νομικές έπτυχες. Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί ευρωβουλευτέ, αγαπητοί συνάδελφοι. Μετά από την παρέμβαση αυτή του συναδέρφου Ρομπέρτο Κάρνε, ο οποίο ε, έβαλε τι βάσει του τι συμβαίνει, του τι ισχύει στο Καθεστώ των υπαλλήλων και των συμβασιούχων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όντω είναι προ όφελο τη υπηρεσία να έχει συμβασιούχου. Σα τα εξήγησε αυτό ο συνάδελφο. Εγώ θα κάνω κάποιε παρατηρήσει από αυτόν που ζήτησε ο αναφέρον. Πρώτον, για την εφαρμογή της οδηγίας. 1989-90 ε, για την ε, ορισμένου χρόνου απασχόληση. Είναι μια οδηγία η οποία πέρασε, εγκρίθηκε και ενσωματώθηκε στις χώρες μέλη. Δεν απευθύνεται στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Έχουμε ένα μηχανισμό βέβαια στο καταστατικό μας που επιτρέπει κάποιες οδηγίες να τις εφαρμόζουμε στο προσωπικό μας. Αλλά αυτό συμβαίνει σε περιορισμένα πλαίσια όταν πρόκειται για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Υπάρχει δηλαδή ήδη αυτός ο περιορισμός. Αυτός ο περιορισμός όμως λίγα μας προσφέρει γιατί ο νομοθέτης που είναι εδώ και το Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και Συμβούλιο λοιπόν, έχουν καλύψει τους υπαλλήλους μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και προστατεύουν βάσει της οδηγίας όλους τους υπαλλήλους. Η οδηγία δηλαδή θέλει να αποφεύγεται ο πολλαπλασιασμός των συμβάσεων και βάσει τρεις προϋποθέσεις, προϋποθέσεις που ακριβώς έχουν σαν στόχο να περιορίσουν την ανανέωση επάπειρο των συμβάσεων αυτών. Και έτσι λοιπόν με εκπλήση που διαβάζω ότι θα έπρεπε να σταματήσει το όριο αυτό των 6 ετών. Ο συνάδελφος το εξήγησε πριν, πήγε από 3 στα 6 χρόνια η περίοδος αυτή, γιατί η οδηγία το λέει ρητά ότι πρέπει να υπάρχει περιορισμό στο χρόνο. Οπότε είτε εφαρμόζεται είτε δεν εφαρμόζεται η οδηγία, πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι εν τη σοφία του, ως οι συνομοθέτες, προέβλεψαν το ίδιο επίπεδο προστασίας όπως θέλαν οι πολίτες. Οπότε σε αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε αυτό. Δεύτερον, η διαφορά ανάμεσα στο μη μόνιμο προσωπικό και το μόνιμο στη χάρτα ποτέ η Επιτροπή δεν αφισβήτησε ότι εφαρμόζεται στους ε, μη μόνιμους όπως και η συνθήκη. Φυσικά, αλλά Μπορεί κάλλιστα να υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα σε ένα σύστημα μονίμων και ένα σύστημα προσωρινών υπαλλήλων που είπε και το δικαστήριο και το επεθύμησε ο συνάδελφος ότι εφόσον υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι που δικαιολογούν τέτοιου είδου απασχόληση, αυτή επιτρέπεται κάλλιστα. Και οι νομοθέτες το προέβλεψαν στο καταστατικό ένα σωρό για τους οποίους μπορεί να υπάρξει αυτή η προσωρινή απασχόληση, κάτι το οποίο αποδέχτηκε πλήρως την ομολογία το δικαστήριο. Οπότε δεν αντιλαμβανόμαστε την αναφορά αυτή, γιατί κάποια στοιχεία της πάνε κατά των όσων αναφέρει η οδηγία, από την άλλη το καταστατικό καλύπτει πλήρως τους συναδέρφους αυτούς και ποτέ το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν την καταδίκασε. Τώρα η βελτίωση που έγινε με τη μεταρρύθμιση του 2013 με την πίεση επίσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν να επιτρέψει μια πασαρέλα, δηλαδή κάποιοι συμβασιούχοι να μπορούν να περάσουν σε μόνιμη απασχόληση. Δεν υπήρχε τέτοια πρόβλεψη νωρίτερα, γιατί δεν είναι εύκολο να γίνει το πέρασμα αυτό, γι' αυτό και λίγοι περνάνε από τη μεθέ στην άλλη. Γιατί, γιατί οι συμβασιούχοι πληρώνονται από τον προπολογισμό. Και το γνωρίζετε όλοι πάρα πολύ καλά. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι υπάρχει ένα συνολικό κονδύλιο που μεταφράζεται σε συμβάσει. Ενώ οι μόνιμοι υπάλληλοι προβλέπονται από τον αριθμό των προσωπικών που προσδιορίζεται αναβαθμό κλπ. Όταν λοιπόν ένα συμβασιούχο πάρει μια μόνιμη θέση, πρέπει να δημιουργηθεί αυτή η θέση. Και αυτές οι θέσεις είναι πολύ περιορισμένες. Είναι ήδη η αρχή του προπολογισμού Εδώ το Κοινοβούλιο δηλαδή και το Συμβούλιο που προσδιορίζουν πόσε θα είναι αυτέ οι θέσει. Οπότε υπάρχει μεν η δυνατότητα αυτή του περάσματος από την Πασαρέλα, αλλά είναι περιορισμένη. Και από εκεί και πέρα όποιο θέλει μπορεί να περάσει διαγωνισμό, έτσι για να γίνει μόνιμος υπάλληλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά ήθελα να σας υπενθυμίσω, αυτά τα νομικά στοιχεία και εδώ ολοκληρώνω την παρέμβασή μου. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, οι συνάδελφοι που θέλουν να συμμετάσχουν στη συζήτηση. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Κύριος Βαλέσα πρώτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, δεν καταλαβαίνω καλά την κατάσταση, γιατί ε, προσπαθούμε να παρακολουθούμε το πώς εξελίσσεται η εργασιακή νομοθεσία στα ε, διάφορα κράτη-μέλη. Και έχουμε τώρα και την Επιτροπή και τους συμβασιούχους υπαλλήλου της και αντιλαμβάνομαι τη διάκριση ανάμεσα στους μονίμους υπαλλήλου και τους συμβασιούχους αλλά υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι συμβασιούχοι υπάλληλοι ε, με ε, ανώτατο όριο ε, περίοδου εργασία 6 ετών στη θέση του, ασχέτω του αν είναι αποτελεσματική ή όχι στην άσκηση των καθηκόντων τους. Δηλαδή πρέπει να τηρείται αυτή η προθεσμία των 6 ετών. Οπότε ποιο είναι το νόημα αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή εκπαιδεύουμε αυτά τα άτομα, επενδύουμε δηλαδή χρόνο και χρήμα στην κατάρτισή του και από εκεί και μετά, μετά από 6 ότι είμαστε υποχρεωμένοι να απολύσουμε αυτά τα άτομα και θα πρέπει να προσλάβουμε νέου συμβασιούχου υπαλλήλου, του οποίου θα πρέπει εκ νέου να καταρτήσουμε. Οπότε, ε, εγώ ε, νομίζω πω θα έπρεπε να παραμείνει ανοιχτή η αν λόγω αναφορά. Θα πρέπει να αναμείνουμε δηλαδή την επόμενη αναθεώρηση ε, του κανονισμού προσωπικού και νομίζω πω θα υπάρξει και μια ακρόαση, αν δεν κάνω λάθο, για τα εργασιακά δικαιώματα το Νοέμβριο, εδώ από την Επιτροπή Αναφορών. Οπότε α αφήσουμε την αναφορά αυτή ανοιχτή και α την βάλουμε στην ημερήσια διάταξη ε, τη ημέρα εκείνη που θα γίνει λόγω ακρόαση. Γιατί δεν κρίνω ικανοποιητική την απάντηση που μα έδωσε η Επιτροπή. Ευχαριστώ. This also never happens, I tell you. Now, Mrs. Ευχαριστούμε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Άσπρουκ για την τόσο ζωντανή παρουσίασή του. Όπως ξέρετε όλες οι ομάδες συμφωνούμε να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά αυτή γιατί για μένα, ιδίω τώρα που έχω ακούσει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν μιλάμε τόσο για μια διεκδίκηση εργασιακή, για παράταση των προθεσμιών που προβλέπεται από μια οδηγία. Πρόκειται για τη συνοχή, τη συνέπεια. Και για μένα δεν υπάρχει συνέπεια ανάμεσα σε αυτά που αμφισβητεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την επισφάλεια της εργασίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γιατί το λέω αυτό. Γιατί υπάρχει αντίφαση σε αυτά που λέτε. Γιατί μιλάτε στην αρχή για προσωρινές συμβάσεις, έτσι, συμβασιούχους, προσωρινούς, που αντικαθιστούν μόνιμους. Με αυτό συμβαίνει. Αν δίνουμε συμβάσεις περιορισμένου χρόνου σε κάποιους, είναι γιατί είναι περιορισμένες οι θέσεις των μονίμων και δεν μπορούμε να έχουμε περισσότερους μονίμους. Αν όμως αυτοί οι άνθρωποι κάνουν μια δουλειά μόνιμη, γιατί να είναι προσωρινή. και είδαμε, όπως το υπενθυμίσατε κι εσείς, ενώ στην αρχή επρόκειτο για έναν πολύ περιορισμένο χρόνο οι συμβάσει αυτές, μετά παρατάθηκε η προθεσμία αυτή. Έφτασε τα έξι χρόνια. Ε, τώρα πείτε μου εσείς τι το προσωρινό έχει μια δουλειά έξι ετών όταν κάποιος κάνει μια πολύ συγκεκριμένη δουλειά για έξι ολόκληρα χρόνια, ε, το προσωρινό είναι αυτό δεν είναι δυνατόν. Έπειτα εσείς μας λέτε ότι ο περιορισμός αυτός, ο χρονικός, τα έξι χρόνια, είναι για εξυπηρέτηση. Γιατί οι συμβασιούχοι δεν πρέπει να χάνουν την επαφή με την έξω αγορά εργασίας. Ναι, αλλά άμα θέλουν αυτοί να δουλέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουν να κάνουν σταδιοδρομία, δεν είναι ότι περνάνε από εδώ να δούνε πώς είναι εδώ τα πράγματα και μετά θέλουν να πάνε αλλού. Όχι, δεν τους εξυπηρετούμε όταν τους περιορίζουμε τις δυνατότητες να απασχοληθούν μονίμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα το στοιχείο κλειδί. Λέτε ότι ένας... Λέτε ότι θέλετε να υπάρχει γεωγραφική ισορροπία ανάμεσα σε μεγάλες και μικρές χώρες. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το κριτήριο. Τι σχέση έχει εδώ με τους συμβασιούχους. Εδώ δεν μιλάμε για τους ανθρώπους που έρχονται από διαφορετικά μέρη και τους βάζουμε στη ζυγαριά. Και για τους διαγωνισμούς λέτε ότι παραμένουν ανοιχτοί και μπορεί οποιοδήποτε να συμμετάσχει. Ναι, αλλά τότε γιατί οι συμβασιούχοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν, αφού λέτε ότι υπάρχουν και ποσοστώσεις πολύ περιορισμένες για αυτούς. Εδώ μιλάμε για μια έκκληση, μια αναφορά που έχει να κάνει με τις βασικές αρχές και την ίση αμοιβή για ίδια εργασία. Κυρίως όμως πρέπει να είμαστε συνεπείς και να μην λέμε ε, μπουρδες από που έρχεται κάποιος και ανάλογα να αποφασίζουμε. Μην λέμε ότι ισχύουν τέτοια πράγματα, δεν συμβαίνει αυτό. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε τις διατάξεις που ισχύουν και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και να μην κρυβόμαστε πίσω από διάφορα άλοθη. Mrs. Βαλίνα. Και κυρία Βαλίνα. Καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ τον αναφέροντα για την τόσο καλή παρουσίαση που μας έκανε, τόσο ξεκάθαρη και τόσο συμπαθητική. Όντως, μας εκπλήσει, μας εκπλήσει που βρισκόμαστε εδώ και ακούμε ότι η ίδια κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που αυτό είναι, έχει 20% συμβασιούχους, που είναι προσωρινοί απασχολούμενοι. Η κατάσταση αυτή είναι ανήκουστη για ένα όργανο μάλιστα το οποίο απαιτεί από όλες τις χώρες μέλη να τηρούν τους κανόνες, τις αρχές, τις αξίες κτλ. Η πρώτη που θα έπρεπε να δίνει το παράδειγμα θα έπρεπε να ήταν η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι εσωτερικοί κανόνες λοιπόν αποκλείουν αθέμητα αλλά αποτελεσματικά τους ίδιους ανθρώπους οι οποίοι έξι χρόνια καταρτίστηκαν, απέκτησαν δεξιότητες, γνώσεις για τη δουλειά τους και μετά δεν μπορούν κάτω από τις ίδιες συνθήκες να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς όπως και οι υπόλοιποι. Οπότε, ούτε εργασιακά ούτε και οικονομικά στέκει, γιατί σκεφτείτε το κόστος κατάρτισης των εργαζόμενων αυτών, αποσβαίνεται με το χρόνο το κόστος αυτό. Και μιλάμε για δημόσιο χρήμα, έτσι. Άρα σπαταλούμε δημόσιο χρήμα με αυτή την τακτική. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν τηρεί μια βασική αρχή που είναι αυτή της μη διάκρισης. Και γι' αυτό το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να μελετήσουμε σε βάθος την υπόθεση, να δούμε πώς μπορούν να αλλάξουν οι διατάξεις που διέπουν ε, τις συνθήκες που ισχύουν για αυτή την κατηγορία υπαλλήλων και κάνω και εγώ την ίδια πρόταση που έκαναν και οι προηγούμενοι, δηλαδή να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά αυτή και να μελετηθεί στην ακρόαση που θα έχουμε το φθινόπωρο για την επισφάλεια των εργαζομένων. Από εκεί πρέπει να αρχίσουμε και εμείς να είμαστε το παράδειγμα. Thank you, Mrs. Ευχαριστούμε κύριε Εύη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τα όσα άκουσα από τους συναδέλφους. Ε, επί το θέμα της αυτής της αναφοράς και ευχαριστώ και τον αναφέροντα ε, που ήρθε εδώ να την παρουσιάσει και την υποστηρίζω, θέλω να το πω καθαρά και από πλευράς μου μεγάλη υποστήριξη για την αναφορά αυτή διότι φέρνει στην επιφάνεια ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που εξακολουθεί να διαπράττεται και από τα ευρωπαϊκά όργανα Πράγματι, οι όροι εργασίας ε, των ε, συμβασιούχων ε, είναι ίδιοι με των μονίμων και μάλιστα αυτοί πολύ συχνά αναλαμβάνουν τεράστιες ευθύνες και πολύ μεγάλο κομμάτι των εργασιών των ευρωπαϊκών όργανων. Είναι λοιπόν θεμέλιος λήθος για τα θεσμικά όργανα και τις εργασίες τους. Και αυτό που συζητάμε τώρα είναι την αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης ε, ε, και ειδικότερα για ανθρώπους που ήδη εκτίθενται σε επισφαλή εργασία και σε, στον κίνδυνο της ανεργίας. Αυτό πρέπει να το διορθώσουμε, να το αποκαταστήσουμε. Αυτό που επηρεάζεται επίσης είναι και το μοντέλο της ε, χρηστής διοίκησης. Διότι, πώς να σα το πω, μου έρχεται να πω ότι είναι σαν να μην υπάρχει πρόθεση να εργαστεί κανείς σωστά προς εξυπηρέτηση των Ευρωπαίων πολιτών ε, κάντα σωστά τη δουλειά μας, τη δουλειά των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων με τρόπο άριστο για τη μέγιστη προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών ε, αν είναι να συνεχίσουμε με αυτό το σύστημα. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπαν οι συνάδελφοι. Η αναφορά αυτή θεωρώ πρέπει να παραμείνει ανοιχτή. Θα μπορούσε να αποτελέσει μια τέλεια ευκαιρία να προσθεθεί στην ημερήσια διάταξη, όπω είπαν και άλλοι συνάδελφοι, τη ε, δημόσιας ακρόασης που θα διοργανώσουμε τον Νοέμβριο. Ακριβώ διότι το ζήτημα πρέπει να συζητηθεί και να επιληθεί το συντομότερο δυνατόν. Δεν έχουμε άλλο χρόνο για χάσιμο, οπότε ευχαριστώ τον αναφέροντα και τους συναδέλφους ε, που θα διατηρήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Κέρτιν Ντάρλινγκ. Σα δώσω ε, συγγνώμη. Ε, ζητώ συγγνώμη στο, από τον αναφέροντα που δεν ήμουν εδώ για να ακούσει την παρουσίασή του γιατί ε, υπήρξε ένα μικρό αυτογενιστικό ατύμα το οποίο είχα. Ε, τώρα, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι την τελευταία εβδομάδα ε, εμεί στο Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο, υιοθετήσαμε ένα ψήμα σε ό,τι αφορά τι επισφαλεί συνθήκε εργασία και νομίζω πω ε, ε, θα πρέπει σε συνέχεια αυτού του ψηφίσματος να καλέσουμε την Επιτροπή να εφαρμόσει στην πράξη τα όσα θεωρητικά ε, υποτίθεται πως υπερασπίζεται. Και βέβαια και εμείς από την πλευρά του Κοινοβουλίου θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε και εγώ υποστηρίζω το να παραμείνει εν λόγω αναφορά ανοιχτή. Και επίσης η ε, ιδέα που έχει ο κ. Βαλέντσα, δηλαδή να προσθεθεί αυτή η αναφορά στην μέση διάταξη της ακρόαση που θα έχουμε τον Νοέμβριο είναι κάτι που υποστηρίζω. Ε, νομίζω πω θα πρέπει να ασκήσουμε πιέσει προκειμένου να υπάρχουν πιο σταθερέ συνθήκε εργασία γενικότερα στην απασχόληση και στι ε, συμβάσει εργασία. Δηλαδή, όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι ε, τέτοια είδου σταθερότητα στην απασχόληση οδηγεί σε πιο υγιή κοινωνία σε ό,τι αφορά δηλαδή την, ψυχοκοινωνική υγεία των εργαζομένων και τι ίδιε τι συνθήκε εργασία. Οπότε θα πρέπει να θεωρήσουμε πω τέτοιου είδου σταθερότητα αποτελεί μια, μια, μικρόθεσμη επένδυση πέραν των άλλων επιχειρητημάτων ότι δηλαδή απολύουν ανθρώπου του οποίου έχουμε εκπαιδεύσει και ούτω καθεξή. Υπάρχει λοιπόν αυτή η διάσταση η οποία μα ε, πιέζει ή μα καλεί να καταπολεμήσουμε κάθε μορφή επισφαλού απασχόληση. Επίση, θα ήθελα να ε, ε, υπενθυμίσω ότι εμείς βρισκόμαστε εδώ ως Επιτροπή Αναφορών στην αιχμή του δόρατος σε ό,τι αφορά αυτές τις πιέσεις. Από το 2009 είχαμε ε, πιέσει για την αναθεώρηση, για παράδειγμα, των κανόνων των ιστορικών διαγωνισμών και δεν θα πρέπει να σταματήσουμε τώρα αυτόν τον αγώνα που έχουμε ξεκινήσει ως Επιτροπή Αναφορών. Θα πρέπει να βρούμε δηλαδή τους τρόπους με τους οποίους θα βελτιώσουμε περισσότερο τις συνδικές εργασία ε, των συμβασιούχων όταν θα έρθει η επόμενη αναθεώρηση ε, του σχετικού κανονισμού. Πάντως, επαναλαμβάνω, όταν λέμε ότι θέλουμε να μην υπάρχει επισφαλή απασχόληση, τότε θα πρέπει να κάνουμε και τα όσα βαγγελιζόμαστε ε, στην πράξη. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρο, κυρία Ντανόκ. Ευχαριστώ. Δεν θα επαναλάβω τα επιχειρήματα που ανέφεραν ε, οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Τα συμμερίζομαι πλήρω και υποστηρίζω ε, αυτή την αναφορά. Γνωρίζουμε ε, πως πάντοτε υπάρχουν αυτά τα προβλήματα όταν γίνονται αναφορές στον ε, ε, χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ειδικότερα δε στο άρθρο 51, όπου αναφέρονται περιορισμοί σε ό,τι αφορά μόνο τις, τα, θέματα που άπτονται των, της αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ένωσης. Εδώ βέβαια έχουμε να κάνουμε πραγματικά με ένα τέτοιο τομέα, δηλαδή τομέα πλήρους ε, αποκλειστικής αμμοδιότητας της Ένωσης και κατά συνέπεια μπορούμε να βασιστούμε στο χάρτη. η δική μου πρόταση θα ήταν ε, καθώς εκπροσωπώ και την Επιτροπή Αναφορών ε, στην Επιτροπή Απασχόλησης και στο σχετικό δίκτυο, η δική μου λοιπόν πρόταση θα ήταν να αποσταλεί ε, εν λόγω αναφορά στην Επιτροπή Απασχόληση. Και εγώ θα ήμουν διατεθειμένη να την παρουσιάσω εκ μέρου μα. Σε ό,τι αφορά τώρα την ακρόαση το Νοέμβριο, ε, δεν είμαι καλά ενημερωμένη. Θα συνδιοργανωθεί με κάποια άλλη Επιτροπή Κοινοβουλευτική. Ε, Πάντω, εάν ναι, θα είναι κοινή δηλαδή αυτή η ακρόαση, καλό θα ήταν η άλλη Επιτροπή να είναι Επιτροπή Απασχόληση. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρο. Ολοκληρώνεται εδώ λοιπόν κατάλογο ε, των συναδέλφων που θέλουν να πάρουν το λόγο, οπότε δίνω και πάλι το λόγο στον κύριο Ασμπρουκ για μια δευτερολογία έως δύο λεπτών. there isn't time, of course. Ναι. Θα μπορούσαμε να απορρίψουμε αν είχαμε το χρόνο τα όσα μας είπε η Επιτροπή, αλλά εδώ θα κάνω μια πρόσκληση Επιτροπή. Ας κάνουμε μια διμερή συζήτηση σε μια ήσυχη αίθουσα συνεδρίασης όπου θα δημοτογραφούμαστε. και εάν δεν δεχτείτε αυτή μου την πρόκληση, τότε θα ε, υπάρξει ένα βίντεο από την πλευρά μου που θα πω φοβάται η Επιτροπή. Ε, Πάντω, αν ρίξει κανεί μια ματιά στο πρώτο άρθρο ε, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ε, πώ μπορείτε, Επιτροπή, να συμβιβάσετε, να συμφιλειώσετε τι πρακτικέ ε, που εφαρμόζετε με την αξιοπρέπεια. Δεν αντιλαμβάνεστε ότι τα άτομα που έχουν επισφαλή απασχόληση δεν είναι πολίτε ε, με, με την πλήρη έννοια. Δεν βλέπετε δηλαδή ότι βρισκόμαστε σε μια ε, φθήνουσα, αν θέλετε, ε, ε, πορεία σε ό,τι αφορά την απασχόληση, ε, όπου δηλαδή κινούμαστε όλο και περισσότερο προς τη δουλεία. αντί όμως τώρα να αναγκάζουμε τους ε, σκλάβους να κοπηλατούν ακόμα πιο γρήγορα, τους ε, πετάμε από το πλοίο. Ε, και βέβαια εδώ τώρα είναι παγιωμένη αυτή η τακτική. Μετά από έξι χρόνια δηλαδή ούτως ή άλλως πετάμε τον ε, σκλάβο από το πλοίο. Ακόμα κι αν έχει γίνει πια ειδικό στην κοπηλασία και έχει μεγάλους μυς. Άρα λοιπόν τόσο για ηθικούς λόγους όσο και για λόγους ρεαλιστικούς σας καλώ να υποστηρίξετε την αναφορά μας και σας παρακαλώ επίσης να διασφαλίσετε ότι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, λέγει δηλαδή, να ενημερωθεί προκειμένου να ενσωματώσει αυτή την αναφορά στην ε, επόμενη αναθεώρηση του κανονισμού του προσωπικού, όπως έγινε άλλωστε και με την αναφορά 192 του 2009. Σας ευχαριστώ, πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα. Σας ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Άρα θα προσπαθήσω εγώ λοιπόν να συνοψίσω τη συζήτηση που έγινε σήμερα εδώ. Ε, αυτό που πιστεύω πως θα πρέπει να κάνουμε είναι να στραφούμε προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί αυτή τη αναφορά. Εγώ συμμετείχα σε εκείνη την επιτροπή όταν έγινε η τελευταία αναθεώρηση και μάλιστα ήμουν ισχυώδη συγκίτρια τη κυρία Ρο Μπέρεν και δεν έχει παρέθει πολλή χρόνο από τότε. Αλλά παρόλα αυτά η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θα έπρεπε να εξετάσει αυτή την αναφορά. Θα μπορούσαμε λοιπόν να το κάνουμε αυτό και θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε το ζήτημα, δηλαδή το θέμα αυτή τη ε, αναφορά στην ακρόαση που θα διοργανώσουμε στι 22 Νοεμβρίου. Αυτά λοιπόν θα κάνουμε σε σχέση με την αναφορά. Προφανώς θα μείνει ανοιχτή η αναφορά. Δεν χρειάζεται να το πούμε καν αυτό. Και αυτά θα κάνουμε. Και βέβαια μπορούμε να αποστείλουμε την αναφορά και στην Επιτροπή Απασχόλησης, αλλά ενημερωτικά και We... Περνάμε λοιπόν στην επόμενη αναφορά. 15-19 σε ό,τι αφορά έργο κατασκευής γραμμής μεταφοράς συνάρτησης υψηλής τάσης στο Fuerteventura. Ε, Γιονένα Καρεσάν ε, Καρμόνα, η, ε, η αναφέρουσα, και της δώσω το λόγο μόλις αποχωρήσουν όσοι το επιθυμούν από την αίθουσα. Now I Ωραία, συνεχίζουμε με το επόμενο θέμα λοιπόν, που είναι η ηλεκτρική γραμμή στην Φουέρτα Βεντούρα. Θα δώσω το λόγο στους αναφέροντες. Παρακαλώ. Γεια σας, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε σημασία και μα δώσετε την ευκαιρία να έρθουμε εδώ σήμερα. Ήρθαμε να ζητήσουμε τη στήριξή σα και τη βοήθειά σα για να στηρίξουμε κι εμεί αυτού που ζουν στην Φορτεβεντούρα και γενικότερα στα Κανάρια όπου πιστεύουμε ότι υπάρχει μια επιχείρηση ηλεκτρισμού, η Red Electrica, που έχει μονοπόλιο, η οποία ε, είναι η μόνη που μπορεί να μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια και να λειτουργήσει το ηλεκτρικό σύστημα. Έχει λοιπόν μονοπόλιο πλήρε όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια σε ολόκληρη την Ισπανία. Κάποιες από τις πρακτικές ε, της Red Electric, αυτής της επιχείρησης ηλεκτρισμού της Ισπανίας, αντιβαίνουν στην νομοθεσία και στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα και σε εκείνα των πολιτών. Θα σας παρουσιάσουμε κάποια παραδείγματα από αυτά που έχουμε στην Φορταβεντούρα και στον Λαθαρότε. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει παρέμβαση αρνητική επιθέσεις βασικά σε ζώνες που περιλαμβάνονται σε οικολογικά δίκτυα όπως το δίκτυο Natura 2000. Επίσης, παρεβιάζεται η χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων που λέει ότι όλοι οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Και τρίτον, εφαρμόζει πρακτικές μονοπωλίου μη ελεγχόμενες που οδηγούν βέβαια σε καταχρήσεις. Η επιχείρηση αυτή ηλεκτρισμού της Ισπανίας έχει διάφορα έργα στα Κανάρια για να μεταφέρει ηλεκτρισμό ε, στα νησιά, κυρίως στην Φορταβατούρα και στο Λανθαρότε που είναι τα μόνα νησιά που συνδέονται ηλεκτρικά. Ε, υπάρχει λοιπόν ένα σχέδιο το οποίο έχει επιπτώσει στο δίκτυο Natura 2000 και στην οδηγία για τα πτηνά. Ε, το πρόγραμμα αυτό λοιπόν επηρεάζει ειδικέ ζώνες διατήρησης, επηρεάζει περιοχές κοινοτικού ενδιαφέροντος και ζώνες ειδικής προστασίας πτηνών. Οι ζώνες αυτές είναι ζώνες στις οποίες ε, βλέπουμε ηλεκτρικές στήλες ύψους πάνω από 50 μέτρα υψηλής ε, τάσης και κάποιους ε, υποσταθμούς ηλεκτρικούς, οι οποίοι ουσιαστικά είναι κάτι τεράστια κτίρια, τεράστια, αν λάβει υπόψη του κανείς το τοπίο και το μέγεθος των νησιών. Οι επιπτώσεις λοιπόν είναι τεράστιες σε ένα τόσο εύθραυστο χώρο όπως είναι ο νησιωτικός και έχουν επιπτώσεις και στην οικονομία και στο περιβάλλον αλλά και στην ευημερία την ίδια των πολιτών. Μέχρι σήμερα έχουμε διαπιστώσει ότι οι επιπτώσεις αυτές οι αρνητικές δύσκολα διορθώνονται. Είτε πρόκειται για την ακτή του Κοραλέχο Αλτοστόν είτε πρόκειται για το Χάμπλε Τελίστ Μοντεχάντια, με έργα τα οποία όπως έχουν σχεδιαστεί τα έργα οδηγούν σε καταστροφές. Με τις πληροφορίες που έχουμε σήμερα μπορούμε να σας πούμε ότι το σχέδιο αυτό της ε, επιχείρησης ηλεκτρισμού της Ισπανίας στην Λανθερότητα και στην Φερτανδούρα τεχνητά έχει κατακαιρματιστεί σε 15 τεχνικά σχέδια τουλάχιστον σε 6 μελέτες ε, αξιολόγησης επιπτώσεων και αυτά έχουν γίνει τελώς τεχνητά γιατί, Γιατί έτσι παράνομα διευκολύνονται οι διοικητικές διαδικασίες, δηλαδή η παροχή άδεια για τα έργα και την μετέπειτα εκμετάλλευσή τους. Οι πραγματικές επιπτώσεις είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθούν και να ληφθούν μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος αποτελεσματικά. Επιπλέον, επίτηδες έχει εμποδιστεί η συμμετοχή των πολιτών στην λήψη αποφάσεων για το περιβάλλον, όπως προβλέπει όμως η κοινωτική νομοθεσία. Τα διάφορα αυτά υποσχέδια είναι σε διαφορετικά σχέδια εξέλιξης, κάτι το οποίο μας δυσκολεύει πάρα πολύ να τα παρακολουθήσουμε. Κάποιες διαδικασίες βρίσκονται μάλιστα και στα δικαστήρια. Άλλες μόλις ξεκινάνε και άλλες διαδικασίες ολοκληρώνονται. Οι πολίτες ε, λοιπόν έχουν ε, αναλάβει δράση κατά της επιχείρησης αυτής ηλεκτρισμού, λέγοντας ότι είναι εντελώς αυθαίρετη η δράση της. Και δεν είναι η πρώτη φορά που η επιχείρηση αυτή οδηγείται σε αυθαίρετες δράσεις με μονοπόλιο των συνδέσεων ηλεκτρισμού της Ισπανίας με άλλες χώρες, είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε εκτός. Επίσης δεν υπάρχει ένας οργανισμός ε, ρυθμισμένος ελεγκτικός στην Ισπανία και αφήνει την επιχείρηση αυτή να μονοπολεί, να χαίρει το μονοπωλίο της. Και οι αποφάσεις ζημιώνουν τους πολίτες. Αυτό το σχέδιο λοιπόν μπορεί να είναι μια νέα περίπτωση κατάχρησης διότι δεν χρησιμοποιεί άλλες εναλλακτικέ λύσεις που θα ήταν αποδοτικές πολύ περισσότερο και οικονομικά και όσον αφορά το περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη το χώρο μέσα στον οποίο εκτελούνται αυτά τα έργα. Γι' αυτό λοιπόν η οργάνωσή μας, η Φορταβετούρα Σωστενίμπλε, βιώσιμη Φορταβετούρα, ζητάμε από βάθους καρδίας να αξιολογήσετε τα έργα αυτά, στο οποίο προχωράει η επιχείρηση ηλεκτρισμού και να λάβετε υπόψη στα συμφέροντα των πολιτών. Μια καλή διαχείριση του ηλεκτρικού συστήματο που να καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες των πολιτών δεν είναι απαραίτητο να ζημιώνει το περιβάλλον, τους πολίτες ή την βιοπικιλότητα σε ένα χώρο που έτσι κι αλλιώς είναι εύθραυστος. Σας ευχαριστώ πολύ όλους που μας επιτρέψατε να έρθουμε και να σας παρουσιάσουμε την αναφορά μας. Ευχαριστούμε πολύ. Με μεγάλη μας χαρά να στραφούμε και στην Κομισιόν για μια απάντηση. Υπήρξε μια γραπτή απάντηση προς εμάς, προς τη γραμματεία που έφτασε την Κυριακή. Δεν την έχουμε στείλει ακόμα όμως σε κανέναν. Θα ήθελαμε τώρα να ακούσουμε τις δικές σας εξηγήσεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ η οδηγία Habitat προβλέπει ότι οποιαδήποτε ε, έργο μπορεί να έχει επιπτώσεις στην προστασία ε, περιοχών ε, που υπάγονται στο Natura 2020 όπως οι περιοχές ειδικής προστασίας θα πρέπει να υποβάλλονται σε ειδικό έλεγχο με βάση τους στόχους διατήρησης της εν λόγω περιοχής και οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να δώσουν τη σύμφωνη γνώμη τους για το εν λόγω έργο μόνο εφόσον βεβαιωθούν ότι δεν έχει ανητικό αντίκτυπο σε ό,τι αφορά την εν λόγω περιοχή. Σε διαφορετική περίπτωση το έργο μπορεί να εκτελεστεί μόνο για λόγους ανωτέρας βίας δηλαδή ε, ε, ξέχοντος δημοσίου συμφέροντος ε, και επειδή δεν υπάρχουν εναλλακτικέ λύσεις και πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται συμπληρωματικά μέτρα τα οποία θα διασφαλίσουν την γενικότερη συμμόρφωση με τα όσα προβλέπονται στο πλαίσιο του δικτύου Natura. Η Επιτροπή λοιπόν υπενθυμίζει ότι το 2015 οι αρμόδιες περιφερειακές αρχές έδωσαν μια προσωρινή έγκριση σε ό,τι αφορά τα τρία έργα κατώ των οποίων αναφέρουσα προσφέρει. Έχοντας προβεί στις σχετικέ διαδικασίες, για παράδειγμα, ε, και δημόσια διαβούλευση. Επίσης, η απόφαση για την έγκριση αυτού του έργου, για γραμμή δηλαδή ε, υψηλή τάσης, έχει αποτελέσει το αντικείμενο ε, προσφυγής από τις ε, περιφερειακές αρχές της Φόρτε Βεντούρα ενώπιον των δικαστηρίων. Ε, και στις αρχές του 2017 το ανώτατο περιφερειακό δικαστήριο εξέδωσε μία προσωρινή εντολή για την αναστολή δηλαδή των εργασιών στο έργο προκειμένου να αποφευχθεί άμεσος περιβαλλοντικός αντίκτυπος. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι τα κράτη-μέλη έχουν την κύρια ευθύνη σε ό,τι αφορά την εφαρμογή ε, και την σωστή εφαρμογή της Ευρωπα... ενωσιακής νομοθεσίας διασφαλίσοντας και την κατάλληλη δικαστική προστασία δηλαδή και ε, τα ε, επαρκή μέσα προσφυγής προκειμένου να είναι δυνατόν τα εθνικά μέτρα να συμμορφώνονται με την ενωσιακή νομοθεσία. Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση που αναφέρεται σε αυτήν εδώ την αναφορά, η ε, έγκριση λοιπόν αυτή που δόθηκε για την εκτέλεση του έργου ακόμα ε, εκρεμεί ενώπιον των Ισπανικών δικαστηρίων. Οπότε η Επιτροπή ε, σε αυτή τη φάση δεν επιθυμεί να παρέμβει στην λόγω περίπτωση. Ευχαριστώ. Λέει η Πρόεδρος, ο λόγος στους συναδέλφου, η κυρία Βαλίνα. Καλημέρα και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα την αναφέρουσα για την παρουσία της αλλά και τους διάφορους συλλόγους που προστατεύουν το περιβάλλον που μας ενημέρωσαν για τους κινδύνους από τα σχέδια της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού της Ισπανίας. Εμείς από την Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά ήμασταν ανέκαθεν κατά αυτού του προγράμματος, γιατί θεωρούμε ότι πρόκειται για κατάχρηση που γίνεται από τις αρχές των Καναρίων Ίσων, γιατί παραβιάζονται διάφορες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως πολύ καλά μας ε, τα είπε η παρουσίαση. Πρώτα απ' όλα οδηγίες που έχουν να κάνουν αντίκτυπο στο περιβάλλον, επιπτώσεις ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών έργων επί του περιβάλλοντος, οδηγία πτηνών, οικοτόπων, ενημέρωσης του κοινού κλπ. Ο κατάλογος είναι πραγματικά μακρύς δυστυχώς. Θα ήθελα λοιπόν να επενθυμίσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί πάντα τις ίδιες απαντήσεις μας δίνουν ότι το ανώτατο δικαστήριο των Καναρίων Ίσων σταμάτησε το έργο ακριβώς εξαιτίας της αρχής της πρόληψης. Και εδώ ποτέ δεν χρησιμοποιείται αυτή η αρχή. Θα έπρεπε σε μερικές περιπτώσεις κατά προτεραιότητα να χρησιμοποιείται αυτή η αρχή, γιατί όταν έχει γίνει ζημιά είναι αδύνατο να διορθωθεί μετά. Η κυβέρνηση λοιπόν, και πρέπει να σας πω ότι η κυβέρνηση των Καναρίων Ίσων έδωσε την άδεια αυτή μέσω μιας περίεργης διαδικασίας που έχει να κάνει με τις αρμοδιότητες του Δήμου, της Περιφέρειας. Το Νότοτο Δικαστήριο λέει ότι υπάρχουν ενδείξεις για παρανομίες. Ένα άλλο παράδειγμα νομοθεσίας ε, à la είναι αυτή και έχουμε κι άλλες. Το λιμάνι του Κατρανίγε, με τον νόμο για τα πράσινα νησιά. Είναι πολλά που έχουμε ήδη συζητήσει και θα συνεχίσουμε να τα συζητούμε εδώ στην Επιτροπή μας. Τώρα λοιπόν η κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων και της Φορτανοπούρα έφερε τη διαβούλευση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δυνατότητα να υπάρξει ζημιά στην ε, ζώνη προστασίας των πτηνών. Κοιτάξτε, ε, ακούγεται αστείο, αλλά Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο θα καταστρέψει το περιβάλλον και την Πανίδα και τη Φλωρίδα, διάφορα είδη και πτηνά και μάλιστα ανεπιστρεπτή. Άρα δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Εδώ δεν μιλάμε μόνο για την ηλεκτρική γραμμή από το λιμάνι Ροσάριο μέχρι το Γκραν Ταραχάλ. Το σχέδιο αυτό επίτηδες κατακαιρματίστηκε σε τρία κομμάτια. Επίτηδες για να αποφευθούν οι συνέπειες επί του περιβάλλοντος στη διαδικασία. Πρώτα απ' όλα από το Ρωσάριο μέχρι το Λίβα και από το Καλαχάρα μέχρι τη Βλάνκας και οι επιπτώσεις δεν πρέπει να αξιολογούνται ε, κατά τμήματα, αλλά συνολικά. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να συνειδητοποιήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς εδώ στην Επιτροπή μας τη μεγάλη καταστροφή. Σας είπα το ίδιο το δικαστήριο και μάλιστα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Σεπτέμβριο του 2004 καταδίκασε την Ισπανία. Και δεν υπάρχει και κανένας λόγος, δεν υπάρχει κανένα συμφέρον για τον κόσμο. Είναι ιδιωτικό το συμφέρον. Δεν είναι ανάγκη το έργο αυτό για ε, το νησί. Και τα μέτρα, τα διορθωτικά τα οποία λαμβάνονται είναι πολύ μερικά και δεν φτάνουν. Για άλλη μια φορά έχουμε να κάνουμε με την ενέργεια και πρόκειται για μια επιχείρηση τελικά ιδιωτικού δικαίου που θα ζημιώσει το περιβάλλον μια τόσο έφραστης περιοχής όπως είναι τα Κανάρια. Γι' αυτό και θέλω να ληφθεί υπόψη η αρχή της πρόληψης για να μην γίνει ζημιά που δεν διορθώνεται στη συνέχεια σε αυτόν τον έθραυστο χώρο που είναι το νησί και να στείλουμε επιστολή στις αυτόνομες αρχές των Καναρίων νησών εκφράζοντας την ανησυχία μας για τις αρνητικές επιπτώσεις επί του δικτύου Natura 2000 και για τον κατακαιρματισμό του προγράμματος που δεν εκτιμά σωστά τη ζημιά που θα γίνει στο περιβάλλον. και να το στείλουμε το θέμα και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για να το μελετήσει, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Thank you very much, uh, Mr. Lopez Aguilar. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λόπες Αγγία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πράγματι δεν είναι η πρώτη φορά που τέτοια θέματα για το περιβάλλον τόσο ευαίσθητα φτάνουν στην Επιτροπή μας από την αυτόνομη περιφέρεια των Καναρίων Νήσων. Όπως ξέρετε υπάρχουν αυτόνομες περιφέρειες και κάθε περιφέρεια έχει το δικό της κοινοβούλιο, τη δικιά της κυβέρνηση και το δικό της δικαστήριο. Οπότε καλωσορίζουμε και ευχαριστούμε εδώ την αναφέρουσα από τα Κανάρια που ήρθε και κυρίως επειδή είναι από την Φορτεναβεντούρα και ευχαριστούμε που μας παρουσίασε την υπόθεσή της. Εκείνη μας ευχαρίστησε, αλλά είναι δικιά μας υποχρέωση να την ακούμε. Εκ μέρους λοιπόν των σοσιαλιστών θέλω να συμφωνήσω με την αναφορά και να ζητήσω επίσης να διατηρηθεί ανοιχτή εδώ στην Επιτροπή Αναφορών Να μην ανοιχτή λοιπόν η αναφορά μέχρι να διευκρινιστεί πλήρως το θέμα της ζημιάς στο περιβάλλον που έχει τεράστια σημασία για μας. Τα εξήγησε πολύ καλά, πρόκειται για μια εταιρεία ιδιαίτερα ισχυρή που έχει ολιγοπόλιο για τον ηλεκτρισμό στην Ισπανία και που προβλέπει να φτιάξει στη φορταφετούρα ε, γραμμές υψηλής τάσης. Η Φερταβεντούρα, όπως όλα τα νησιά στα Κανάρια, ε, διαθέτουν ε, πολλές ειδικέ περιοχές προστατευμένες για τα πτηνά, ΣΕΚ, ΠΕΚ και άλλες, οι οποίες κινδυνεύουν να καταστραφούν, άρα να καταστραφούν σπάνια είδη, προστατευόμενα είδη, όπως διάφορα τέτοια πτηνά από αυτά τα καλώδια υψηλής Επιμένω για το Natura 2000 και θα έπρεπε πρώτα να ερευνήσουμε σε βάθος τις περιβαλλοντικές ε, επιπτώσεις βάσει του άρθρου 6 της Οδηγίας για τα Απτινά να απαιτήσουμε μέτρα τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται αυτή τη στιγμή από την εταιρεία Red Electrica. Γιατί ό,τι μέτρα έχει πάρει μέχρι τώρα, όπως επίσης και οι αρχές αντισταθμιστικά, δεν φτάνουν. Το έργο θα καταστρέψει τις λίμνες. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποφύγουμε την καταστροφή των προστατευμένων ειδών με εναλλακτικά μέτρα να ξέρουμε ότι δεν είναι αλήθεια πως είναι αναγκαίο αυτό το μέτρο. Θα μπορούσε υπόγεια να μπουν οι γραμμές αυτές υψηλής τάσης. Αλλά αποκλείστηκε αυτό και καθαρά οικονομικούς λόγους, όχι οικολογικούς ή περιβαλλοντικούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ξέρω κατά πόσο εξέτασε τις εναλλακτικές λύσεις πριν εγκρίνει αυτό το σχέδιο. όσα προβλέπονται στην οδηγία του 2011-92 για τη συμμετοχή των πολιτών σαν βασικό στοιχείο ελέγχου της διοίκησης για να ε, μην υπάρχουν ιδιωτικά συμφέροντα δεν ξέρω αν όλα αυτά τα παρακολούθησε. Πάντως, πρέπει να στείλουμε επιστολή, όπως σας είπα, στις αρχές της περιοχής και να ζητήσουμε το, αυτό το έκανε μάλλον το Κοινοβούλιο των Καναρίων ε, Νήσων με θετική ψήφα των σοσιαλιστών να σταματήσουν τα έργα. Εγκρίθηκε επίσης πρόταση τον Φεβρουάριο νόμος για να ζητήσει να μπουν υπόγεια τα καλώδια αυτά. Η εγκατάσταση δηλαδή είναι υπόγεια Οπότε, εδώ πρέπει να τονίσουμε πόσο μεγάλη σημασία έχουν οι διατάξεις και οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του περιβάλλοντος και των προστατευόμενων ειδών, των πτηνών και η μεγάλη ζημιά που θα πλήξει έθραυστα ήδη και ότι από το έργο αυτό η απειλή είναι τεράστια για όλα αυτά τα είδη. Συνεπώς, συμφωνώ με την αναφορά, ζητώ να παραμείνει ανοιχτή μέχρι να διευκρινίσει πλήρως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι παραβιάσεις γίνονται και τι ζημιά κινδυνεύει να γίνει στα προστατευόμενα αυτά είδη. Ευχαριστούμε για αυτή την πραγματικά μακρά σας παρέμβαση, ο κύριος Κάθε φορά που εμφανίζονται τέτοιες περιπτώσεις και εμφανίζονται πολλές στην Επιτροπή μας, σκέφτομαι ότι υπάρχουν κάποια κριτήρια που πρέπει να λαμβάνουμε πάντα υπόψη, γιατί βέβαια δεν είναι δυνατόν να πετύχουμε την ισότητα αν δεν λάβουμε υπόψη μας τις ιδιαιτερότητες. Στην συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν υπάρχουν δύο πολύ σημαντικά στοιχεία. Το ένα είναι ότι πρόκειται για νησιά και το δεύτερο είναι το μονοπόλιο της επιχείρησης ηλεκτρισμού. Αν λοιπόν αυτά τα δύο τα συνδυάσουμε, ο νησιωτικός χαρακτήρας έτσι και αλλιώς γεωγραφικά αποτελεί μια δυναμία. Έτσι. Αν αυτό λοιπόν το συνδέσουμε με το μονοπόλιο, φτάνουμε σε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, όπως είπε και συνάδελφος, που απαιτεί την αρχή της προφύλαξης. Είναι λοιπόν δυσανάλογο το σχέδιο αυτό το οποίο προβλέπεται για τα νησιά. Και εγώ, ξέρω κάθε φορά η Επιτροπή τα ίδια μας λέει, είναι θέμα χωρών μελών. Ναι, αλλά αν το περιβάλλον, και εγώ βέβαια εντάξει είμαι στην ομάδα των πρασίνων, αν λοιπόν το περιβάλλον δεν είναι ευρωπαϊκό ζήτημα, ε τότε πείτε μου ποιο είναι το ευρωπαϊκό ζήτημα. Συνεπώ, πρέπει να παρεμβαίνουμε σε θέματα περιβάλλοντος ακριβώ γιατί είναι ευρωπαϊκά. Και δύο ακόμα θέματα. Το ένα, να παραμείνει ανοιχτή, βέβαια, η αναφορά αυτή, γιατί υπάρχουν εναλλακτικέ λύσεις, όπως είπε και ο Χαν Φερνάντο, ο Και γιατί υπάρχουν αποφάσεις, όχι πάντα δικαστικέ, αλλά και νοβουλευτικές υπάρχουν από τη χώρα και είναι σημαντικές και γιατί όπως πάντα σε περιπτώσεις μονοπωλίων, έτσι και εδώ, πάρθηκε η απόφαση κατακαιρματισμού του προγράμματος. Άρα μένουν στην πάντα και ξεφεύγουν κάποια ζητήματα τα οποία δεν θα ξέφευγαν αν δεν είχε προκύψει αυτός ο κατακαιρματισμός. Γι' αυτό λοιπόν απαιτώ και εγώ την προφύλαξη και την προτεραιότητα. Η Ρώσα τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Σύμφωνο με όσα είπαν οι συνάδελφοι μέχρι τώρα. Όταν ε, ετοιμάζεται ένα τέτοιο σχέδιο και τώρα χωρίστηκε σε τρία κομμάτια, αυτά τα 14 υπό τμήματα. Όπως είπαμε εδώ, το σχέδιο αυτό θέτει σε κίνδυνο την προστασία των ειδών. Οπότε και εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να τηρεί την νομιμότητα πάνω απ' όλα. Και η Επιτροπή δεν μας απάντησε. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια υπόθεση που σαφώς και πρέπει να μείνει ανοιχτή για να βεβαιωθούμε ότι τηρείται η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο Άγγελες. Καλό θα ήταν να τηρούμε αυτή την αρχή της προφύλαξης, δηλαδή να ξέρουμε εκ των προτέρων αν τηρεί την νομοθεσία, γιατί όταν έχει γίνει ήδη το έργο είναι πολύ αργά. να υπάρχει μια στρατηγική ώστε πριν αρχίζουν τέτοια έργα να μπορούμε να τα σταματήσουμε και να ξέρουμε κατά πόσο τηρείται η νομοθεσία ή όχι, ακόμα και αν τα δικαστήρια από τη δικιά του στην πλευρά παράλληλα κάνουν την δουλειά τους. Ωραία, δεν έχω άλλον ομιλητή στον κατάλογο ομιλητών, οπότε θα δώσω το λόγο και πάλι στην αναφέρουσα δύο λεπτά παρακαλώ για να συνοψίσετε τις εντυπώσεις σας και τι επιθυμείτε εσείς για τη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Επειδή υπάρχει αυτός ο κατακαιρματισμός στο σχέδιο και χρονικά το κάθε τμήμα βρίσκεται σε διαφορετικό στάδιο, στην πραγματικότητα υπάρχουν έξι κομμάτια, όχι τρία και συνεχίζονται οι δικαιωτικές αρχές του Λανθαρότε τον Ιανουάριο εξέτασε κάποια. Δεν ξέρουμε πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Ο κατακαιρματισμός αυτός ε, έχει σαν αποτέλεσμα ότι και η προσφυγή στο δικαστήριο πρέπει να γίνει ανά κομμάτι. Άρα η οργάνωσή μας δεν μπορεί ουσιαστικά να προσφύγει στο δικαστήριο για όλα αυτά τα κομμάτια. Και αυτό μας ε, θλίβει. Ούτε πληροφορίες αρκετές έχουμε με την ε, χρονική συνέχεια και τον κατακαιρματισμό έχουμε πρόβλημα. Αυτός ο κατακαιρματισμός, το ότι το κάθε τεχνικό κομμάτι του σχεδίου πρέπει να πηγαίνει στα δικαστήρια, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι. Τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ όλους όσοι πήρατε το λόγο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σύνολό του. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε που δώσατε τόσο χρόνο για ένα θέμα που είναι για όλους μας πάρα πολύ σημαντικό. Ωραία, ας προσπαθήσουμε τώρα να κλείσουμε και φυσικά θα κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά, αυτό είναι αυτονόητο. Και πιστεύω επίσης ότι επειδή όπως είπε ήδη η Κομισιόν η υπόθεση αυτή είναι η δράση που αποτελεί ένσταση για την έγκριση του έργου ακόμη εκκρεμή. Γι' αυτό η Κομισιόν δεν μπορεί να αναλάβει δράση. Οπότε εμείς πρέπει να το παρακολουθούμε. Οπότε προτείνουμε να στείλουμε μια επιστολή στις ε, περιφερειακές αρχές όπου θα επισημαίνουμε το πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό και επίσης θα πρέπει να παρακολουθούμε ε, διατηρώντας έτσι την αναφορά ανοιχτή για να επανέλθουμε αργότερα. λέγοντας πολύ σαφώς ότι είναι κάτι που εμείς θα παρακολουθούμε. Και ελπίζουμε ότι η απόφαση που θα ληφθεί θα είναι η σωστή θα στείλουμε τις πληροφορίες ενημερωτικά και στην ε, Επιτροπή ΕΜΒΗ. Ναι, συμφωνείτε για όλα αυτά. Ωραία, ευχαριστούμε. Ε, ευχαριστούμε και πάλι που ήρθατε εδώ. Το σημείο 15 αναβλήθηκε για τον Οκτώβριο. Το σημείο 16. Αυτό θα δούμε τώρα. Αναφορά 1432 σχετικά με το έργο Πασάντε την Πολόνια. Η αναφέρουσα βρίσκεται εδώ. Καλωσορίσατε στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Ο κύριος Λούκα Τασινάρη, εσείς εκπροσωπείτε την αναφέρουσα, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύρια Πρόεδρε, αξιότιμη ε, βουλευτές. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω την αναφορά κατά του Πασάντα της Μπολόνια, ενό αστικού αυτοκινητοδρόμου πλάτους 50 μέτρων, μήκους 13 χιλιόμετρων που διαχειρίζεται η εταιρεία Autostrade per SPA που θα περνάει από γειτονιέ ε, με ε, πυκνούς κατοίκους και η διαπλάτηση κατά 14 μέτρα όπως προβλέπεται αυτή τη στιγμή θα μειώσει ακόμη περισσότερο τις αποστάσεις από τις κατοικίες. Στο Πασάντε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα κινούνται 180.000 οχήματα την ημέρα, 65 εκατομμύρια ετησίως σε απόσταση 10 μέτρων από τα σπίτια, κάτι τελείως παράλογο. Η Μπολόνια βρίσκεται στο κέντρο της ε, κοιλάδας του ε, πάδου μια περιοχή που είναι από τι πιο μολυσμένε στην Ευρώπη. Στου πρώτου μέρε του 2017 καταγράφηκαν 24 υπερβάσει των επιπέδων μικροσωματιδίων και 15 υπερβάσει των επιπέδων όζοντο ε, με όρια μερικές φορές πενταπλάσια από τα νόμιμα. Το διοξίδιο του αζότου είναι σε επίπεδα απαράδεκτα. Αυτοί οι ρήποι εξαρτώνται από την κίνηση των οχημάτων και επηρεάζουν σημαντικά και αρνητικά την ε, δημοσία υγεία το, να διαπλατηνθεί η, ο αυτοκινητόδρομος αυτό σημαίνει ότι ε, ε, επιδεινώνονται οι ζημιές ε, προς την υγεία. Αυτό δεν είναι λογικό και αντίκειται στις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην αναφορά θα βρείτε τις αιτίε που μας τεκμηρώνουν ότι πρόκειται για ένα άχρηστο έργο που δεν θα επιλύσει το πρόβλημα της κίνησης, που δημιουργεί προβλήματα, επιδεινώνει την περιβαλλοντική ε, κατάσταση και είναι ένα έργο αναχρονιστικό διότι η τάση σε όλο τον κόσμο, στο Σαν Φρανσίσκο, στο Αμβούργο, στη Λιόν, στη Μαδρίτη είναι η καταστροφή ε, των ε, αστικών αυτοκινητών δρόμων και όχι η διαπλάτησή του. Είναι απαράδεκτο λοιπόν στην Πολόνια, την πόλη που φιλοξένησε τη διάσκεψη για το περιβάλλον των G7 και που είναι υποψήφια ε, πράσινη πρωτεύουσα ευρωπαϊκή για το 2019 να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση επηρεάζοντας την υγεία χιλιάδων πολιτών. Το έργο αυτό συζητήθηκε σε μια δημόσια διαβούλευση που δεν έχει να κάνει δεν έχει καμία σχέση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες ε, που ορίζονται ε, και από την σύμβαση του Όρχους. Ε, ήταν μια απλή προπαγάνδα αυτή η δημόσια διαβούλευση για μια απόφαση που έχει ήδη ληφθεί από την κυβέρνηση και από τις τοπικές αρχές χωρίς να προσφέρει καμία αναλλακτική. Φανταστείτε ότι ακόμα και η μηδενική επιλογή, δηλαδή η επιλογή του να μην γίνει το έργο, δεν υπήρχε στις συζητήσεις. Η ελληπής ε, συμμετοχή βάθινε το ρήγμα, τη ρήξη, την κοινωνική και πολιτική ε, η επιλογή τώρα αυτή του Πασάτε την Πολόνια έχει ε, μεγεθύνει τη ρήξη και αυτό δεν είναι σωστό. Θα περνάει, όπως είπαμε, από περιοχές ε, όπου ζουν 90.000 από τους 390.000 κατοίκους της Μπολόνια και οι ζημιές στο περιβάλλον και στην υγεία θα είναι τεράστιες με κατάφορη παραβίαση εδώ τη ίσης ε, κατανομής των περιβαλλοντικών κινδύνων. Η Ιταλία εδώ και χρόνια βρίσκεται σε μια διαδικασία παραβάση λόγω ελλειπούς αντιμετώπισης της ε, ατμοσφαιρικής ρήπανσης με μια πολιτική μεταφορών επικεντρωμένη στα αυτοκίνητα ε, που αγνοεί τις εκκλήσεις της Ευρώπης για εναλλακτικές βιώσιμες μεταφορές δίνοντας προτεραιότητα στους σιδηροδρόμους, τα ποδήλατα και ε, τους πεζόδρομους. Ε, στην Εμίλια Ρωμάνια λοιπόν το περιφερειακό σχέδιο για τις μεταφορές προβλέπει 12 δισεκατομμύρια επενδύσεων, 7,5 των οποίων προορίζονται για νέους αυτοκινητοδρόμους, κομμάτι των οποίων είναι και το Πασάντα την Πολόνια, το οποίο αποτελεί εμπεγμό των ευρωπαϊκών οργάνων. Το αίτημά μας προς την Ιταλική κυβέρνηση είναι να παραιτηθεί από αυτό το έργο που είναι επιβλαβές για τους πολίτες και να εφαρμόσει επίσης επιτέλους μια πολιτική μεταφορών που θα προστατεύει το περιβάλλον και την υγεία ε, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Προς την Κομισιόν ζητάμε να εγκρίνει αυτή την αναφορά ως ένα πρώτο βήμα μιας διαδικασίας που θα βοηθήσει ε, να αντιμετωπιστούν ε, αυτές οι υποθέσεις βιώσιμων μεταφορών και στην Ιταλία με τη συμμετοχή των πολιτών. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω η Επιτροπή να υιοθετήσει διάφορες πρωτοβουλίες κατά της Ιταλικής κυβέρνησης ώστε να μην γίνει αυτή η διαπλάτευση του Πασάντε την Πολόνια. Επίσης θα ήθελα ε, κατά της Ιταλικής κυβέρνησης να υπάρξει μια διαδικασία παραβάση του δικαίου της Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει τώρα η Κομισιόν και πρέπει να σας πω ότι η αναφορά είναι πολύ πρόσφατη. Έγινε παραδεκτή 12 Απριλίου μόλις και μετά τη στείλαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ακόμη δεν έχουμε λάβει γραπτή απάντηση διότι είναι πάρα πολύ πρόσφατη αλλά την διεκπαιρεώσαμε με την διαδικασία κατεπήγοντος μετά από έτοιμα από μια πολιτική ομάδα. Γι' αυτό το λόγο έγινε αυτό. Οπότε μην έχετε την αίσθηση ότι δεν έχουμε τις σωστές πληροφορίες, απλά έχουμε ε, ακολουθήσει τη διαδικασία κατεπήγοντος. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Η δική μας ανακοίνωση η αφορά α, καταρχήν ε, το περιβάλλον και από την άλλη πλευρά αφορά τις δημόσιες συμβάσεις. Καταρχήν σε ό,τι αφορά την πρώτη πτυχή, τα ε, ε, κράτη-μέλη είναι τα κυρίω αρμόδια για την εφαρμογή τη ενωσιακή νομοθεσία. Κατά συνέπεια, επαφίεται στι εθνικέ αρχέ να αξιολογούν ε, τον αντίκτυπο, τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο σε όλε τι διαστάσει, δηλαδή ατμοσφαιρική ρήπανση, των εδαφών, των υδάτων και κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία σε σχέση με τέτοια έργα. Άρα λοιπόν αυτέ οι διαστάσει θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντω υπόψη στο πλαίσιο τη διαδικασία EIA προτού δοθεί η έγκριση για την ε, περαιτέρω ανάπτυξη Επίσης η εναλλακτική του να μην λάβει χώρα κανένα έργο θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη και επίσης θα πρέπει να γίνεται ε, και υποβολή των σχετικών ε, σχεδίων στο κοινό, στο πλαίσιο δηλαδή της δημόσιας διαβούλευσης. Με βάση τα όσα έχουμε στη διάθεσή μας, ε, η διαδικασία που ακολουθήθηκε, η διαδικασία ΙΑΕ e δηλαδή, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο έργο, τρέχει ακόμα. Βρίσκεται δηλαδή σε αυτή τη χρονική στιγμή στη φάση της τεχνικής αξιολόγησης, ενώ η δημόσια διαβούλευση έλαβε χώρα από τις 10 Ιανουαρίου στις 13 Μαρτίου του 2017. Η αναφέρουσα υπέβαλε κάποιες παρατηρήσεις τον ε, Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2017. Ενώ από εκεί και μετά τα έργα τα οποία εμπίπτουν ε, στην, ε, στο πεδίο εφαρμογής η ΑΕ, για παράδειγμα, οι ε, μεταφορές ε, ε, μικρών αποστάσεων και οι μικρές τροποποιήσεις που γίνονται σχετικά δίκτυα χρήζουν περιβαλλοντικής αξιολόγησης αντικτύπου μόνο στις περιπτώσεις εκείνες όπου τα κράτη-μέλη θεωρούν πως μπορεί πράγματι να υπάρχει σημαντικός περιβαλλοντικός αντικτύπος. Κατά την διεξαγωγή λοιπόν τέτοιου είδους ε, εποπτεία, αν θέλετε ή παρακολούθηση ε, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους και τους κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία. Με βάση λοιπόν τις πληροφορίες που διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή δεν κατάφερε να ε, εντοπίσει ότι πρώτον δεν έλαβε χώρα κάποια τέτοια παρακολούθηση ή ότι δεν υπήρχε ότι υπήρχε μια βούληση προς το αντίθετο από την πλευρά του κράτους μέλους, ούτε από την άλλη πλευρά δεν υπήρξε ε, κάποια άλλη αρνητική απόφαση. Σε ό,τι αφορά ε, γενικά την οδηγία SCA προβλέπεται ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ε, προτού ξεκινήσει το έργο να εντοπίζουν τους κινδύνους και θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της διαμόρφωσης διαβούλευσης. Πράγμα όμως το οποίο πάντα περιμένει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Επίσης, τα πορίσματα αυτά της διαδικασίας, δηλαδή παρακολούθηση αξιολόγηση στο πλαίσιο της οδηγίας SEA θα πρέπει να καθιστάται δημόσια διαθέσιμα. Τώρα, ε, ε, η οδηγία 2002 του 39 σε ό,τι αφορά την ατμοσφαιρική ρήπανση και τον ε, θόρυβο δεν θέτει συγκεκριμένα όρια σε ό,τι αφορά τον θόρυβο από το του δρόμου. Πάντω, με βάση τα δεδομένα που έχουμε λάβει, με βάση το, τα όρια PM10 e και άλλα, υπάρχει μια θετική εξέλιξη στην Πολωνία τα τελευταία έτη. Επίση, η οδηγία 2008 του 50 δεν προβλέπει συγκεκριμένα όρια, ανώτατε έτοιμε σε ό,τι αφορά τα επίπεδα όζοντο. Επίση, η Επιτροπή δεν ήταν σε θέση να εντοπίσει στοιχεία που θα ε, παρέπεμπαν στην ε, παραβίαση του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων ή ε, των άρθρων της Σύμβασης ε, των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της, των Ηνωμένων Εθνών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις δημόσιες σύμβασεις, η αναφέρουσα αναφέρει ότι με βάση την πολιτική συμφωνία που στις 15 Απριλίου του 2017 μεταξύ των τοπικών αρχών και της επιχείρησης του αναδόχου δηλαδή που έχει αναλάβει την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Α40, κοινοπραξία ουσιαστικά περιλαμβάνει μία σειρά από ε, ε Ιταλικές επιχειρήσεις αποφασίστηκε η κατασκευή δύο ε, ακόμα λωρίδων χωρίς να ε, υπάρξει ε, κανονική διαδικασία διαγωνισμού. Η αναφέρουσα επίσης αναφέρει ότι κάτι τέτοιο βρίσκεται σε άμεση αντίθεση τόσο με την εθνική νομοθεσία όσο και με την ενωσιακή νομοθεσία σε ό,τι αφορά τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις αφού η συγκεκριμένη κοινοπραξία δεν επιλέχθηκε ως ανάδοχος στο πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας διαγωνισμού. Κατά συνέπεια θα ήταν απαραίτητο να ξεκινήσει μια δημόσια διαδικασία, ένας δημόσιος διαγωνισμός προκειμένου άλλε επιχειρήσει οι οποίε δεν συμμετέχουν σε ένα λόγο κοινοπραξία στο συγκεκριμένο όμιλο να μπορέσουν να συμμετάσχουν. Με αυτόν τον τρόπο θα αντισταθμιστεί η απουσία ουσιαστικά της, ε, του ε, ε, ε ανταγωνισμού και το συγκεκριμένο ζήτημα εμπίπτει και στην οδηγία 2014-23 σε ό,τι αφορά τις χωρίσεις. Η 2014-23 και η 2014-25 οδηγίες σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συμβάσεις δεν αφορούν τη συγκεκριμένη περίπτωση σε συγκεκριμένο έργο. Επίση, η Επιτροπή ε, θεωρεί πω η οδηγία σε ό,τι αφορά τι ε, παραχωρήσει δεν προβλέπει κάποια διάταξη που να αναφέρει όπου ένα ε, ε, ανάδοχος ο οποίος δεν έχει ε, επιλεγεί μέσω ε, διαγωνισμού θα πρέπει να διασφαλίσει σε συνέχεια του έργου τον ανταγωνισμό, αυτό το downstream δηλαδή ανταγωνισμό. Ωστόσο, το άρθρο 177 του Κώδικα για τις Δημόσιες Συμβάσεις της Ιταλικής Νομοθεσίας προβλέπει κάτι τέτοιο. Οπότε, εάν αυτή η συμφωνία της 15ης Απριλίου του 2015 ε, προέβλεπε κάτι το οποίο έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 177 του σχετικού κώδικα της Ιταλικής νομοθεσίας θα πρέπει να ε, ληφθούν διορθωτικά μέτρα από τις αρμόδιες διοικητικές Ιταλικές αρχές. Ε, λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη όλα τα παραπάνω και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι τα περισσότερα από τα όσα ε, ζητήματα θέτουν οι αναφέροντες εμπίπτουν στην εθνική αρμοδιότητα τη Ιταλία και λαμβάνοντα υπόψη ότι ήδη έχει κινηθεί διαδικασία ενώπιον των εθνικών Ιταλικών δικαστηρίων η Επιτροπή δεν προτίθεται να αναλάβει περαιτέρω δράση σε σχέση με συγκεκριμένη υπόθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Εύη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους αναφέροντες ε, είναι το χιλιοστό καταραμένο έργο που εντάσσεται στο ευρύτερο σύνολο των διαφόρων καταραμένων έργων που έχουν γίνει μέσα στον χρόνο ε, που υποβαθμίζουν ε, ε, τη φύση, το περιβάλλον, την υγεία σημαντικά για τον πληθυσμό της Μπολόνια. Όπως θυμίσε και ο αναφέρον, οι διάφορες διαδικασίες επαραβάσεις που ενδιαφέρουν την Ιταλία, ειδικότερα όσον αφορά την ποιότητα του αέρα είναι γνωστές. Η κατάσταση πια είναι μόνιμη. Ε, μόνιμη παράβαση, η παραβίαση των ορίων. Αυτό που εμένα με τρομάζει και με ανησυχεί είναι ότι πολλά από τα αιτήματα που απίφθηναν οι πολίτες μέσα στον χρόνο δεν ε, λήφθησαν καθόλου υπόψη. Όπως για παράδειγμα το αίτημα για δεδομένα όσον αφορά τις επιπτώσεις στην υγεία και τα επιδημολογικά δεδομένα που χαρακτηρίζουν την περιοχή αυτή όπου θα γίνει η διαπλάτηση και η βελτίωση του Πασάντα της Μπολόνια. Τα αιτήματα αυτά πέρασαν σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Τα γνώρισαν άπαντες όπως αγνώρισαν ε, και κάθε εναλλακτική λύση για ένα τέτοιο έργο. Ο που θα έπρεπε να είχαν λεφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Κάτι που δεν συνέβη. Μιλάμε λοιπόν για ένα έργο το οποίο προωθείται αποφασιστικά από τις αρχές, τις τοπικές αρχές, χωρίς να υπάρχει οποιοδήποτε περιθώριο λιγμών ή συμμετοχής ε, των πολιτών. Μιλάμε για παραβίαση των κανόνων, των ε, συμφωνιών, των διεθνών συμβάσεων και των ευρωπαϊκών συμβάσεων και σκεφτούμε ειδικότερα τη σύμβαση του Άρχους. Ε, μόλις πέντε εβδομάδες δόθηκαν στους πολίτες για να κάνουν παρατηρήσεις. Αυτό είναι εμπεγμό. Είναι γελίο χρονικό διάστημα. Δεν προλαβαίνει κανεί να ε, κάνει σωστά οποιαδήποτε, να συμμετέχει σωστά ως κοινό. Ε, και ήθελα να σταθώ λίγο σε αυτό. Το έργο αυτό μας το πουλάνε ως βελτίωση της σημερινής κατάστασης και μας διαβεβαιώνουν ότι δεν πρόκειται να επιδεινωθεί η ατμοσφαιρική ρήπανση διότι τα αυτοκίνητα θα κινούνται με σταθερή ταχύτητα και η, η ανανέωση των ε, οχημάτων μέσα στα επόμενα χρόνια θα διασφαλίζει ότι ο αέρας θα είναι καθαρότερος. Εγώ θέλω να πω στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις τοπικές αρχές ότι βρισκόμαστε ε, μην ξεχνάτε, έχουμε το gate, ένα νέο σκάνδαλο που μας λέει ότι πολλά από τα αυτοκίνητα, τα diesel, τα dieselοκίνητα δεν τηρούν τα όρια. Και για να, για να νεωθεί ο στόλο αυτών των αυτοκινήτων θα χρειαστεί μια πενταετία. Οπότε θα συνεχίσουμε να ζούμε σε αυτού του θαλάμου αερίων, όπω έχουν μεταμορφωθεί οι πόλει μα. Ε, θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάποιε λογικέ κινήσει όσον αφορά την κινητικότητα στι πόλει μα. Ε, ε, κινητικότητα που να αφορά τις δημοσίες μεταφορές, τις συγκοινωνίες, ε, ενδεχομένως με ε, κινούμενες με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να βελτιώσουμε τους σιδηροδρόμους, αντί να ευνοούμε μόνο κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα. Εγώ εύχομαι λοιπόν να μην ανοιχτεί αυτή η αναφορά ώστε τα αδιαφανή κομμάτια να εξεταστούν, να τους δοθεί η μέγιστη προσοχή ε, και αν δούμε και το ιστορικό των παλιότερων εργών που εγκαταλείφθηκαν τέλος λόγω διαδικασιών παραβάση ε, Θεωρώ λοιπόν ότι είναι απαραίτητο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Αναφορών να δώσει προσοχή στο θέμα αυτό. Διότι οι απαραβιάσεις μπορεί να είναι πολύ σοβαρέ και επιβαρύνουν το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών της Μπολόνια. Ευχαριστώ. Thank you very much. Mr. Affronte. Ευχαριστώ κύριο Αφρόντε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ πρότεινα στους πολίτες να παρουσιάσουν την αναφορά τους εδώ στην Επιτροπή Αναφορών και χαίρομαι που φτάσαμε μέχρι εδώ. Έχω προετοιμάσει δύο λόγια, αλλά με συγκλώνησε τα όσα είπε η Κομισιόν ουσιαστικά δημιούργησε ένα προπέτασμα καπνού, ε, όπως συχνά βλέπουν οι πολίτες στην ε, Κομισιόν και τα θεσμικά όργανα, ότι βάζουν διάφορους κανόνες, ενώ τα αιτήματά τους είναι πολύ ρητά, πολύ σαφή, πολύ δομημένα. Ε, πολίτες που έρχονται εδώ για να λάβουν κάποιες απαντήσεις πιο καθαρές. Άκουσα από την Κομισιόν ότι οι τάσεις ε, των ρήπων να μειώνονται και αυτό δίνει ελπίδες για την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία των πολιτών. Μιλάμε για μείωση λόγω της οικονομικής κρίσης όπως ξέρουμε όλοι. Γι' αυτό τον λόγο ε, δεν χρειάζεται να κάνουμε άλλη διαπλάτηση αυτού του αυτοκινητοδρόμου και να ε, επιδεινώσουμε τη μόλυνση. Θα μπορούσαμε καμιά φορά να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε αυτό που πάντα συζητάμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή την βιώσιμη κινητικότητα, τις εναλλακτικέ, ε, τη χρήση των συγκοινωνιών, όλα αυτά που συζητάμε διαρκώς εδώ και που με την πρώτη ευκαιρία, με το πρώτο αίτημα των πολιτών τους λέμε ότι ξέρετε στην οδηγία τα έχουμε ρυθμίσει όλα. Αυτό που θέλω να υπογραμμίσω, το έκανε και η συναδελφός μου κυρία Εύη, είναι η συμμετοχή του κοινού, του, των πολιτών δεν είναι μια διατύπωση, όπως συχνά αντιμετωπίζεται δυστυχώς, ε, ειδικότερα στη δική μας χώρα. Δεν είναι απλά ένα ασήμαντο κομματάκι ε, της διαδικασίας. Ε, πρέπει να συμμετέχουν, πρέπει να τους ακούμε τους πολίτες. Δεν είναι απλά για να, να το κάνουμε για να λέμε ότι το κάναμε. Δεν μπορεί να αποτελεί ένα εργαλείο, όπως είπε ε, οι αναφέροντες ε, δεν μπορεί να είναι ένα εργαλείο προπαγάνδας πρέπει να είναι ένα εργαλείο ακρόασης και ξέρουμε ότι αυτό δεν συνέβη οι διαβουλεύσεις δήρξαν ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα διοργανώθηκε αυτή η δημόσια συνάντηση όπου στην πραγματικότητα και εδώ πραγματικά χάνουμε το νόημα της ε, συμμετοχής των πολιτών δεν είναι θέμα ενημέρωσης το θέμα ήταν να τους ακούσουμε και εμείς όχι απλά να τους ενημερώσουμε εμείς και αυτό μαζί με όλα τα υπόλοιπα που ακούσαμε εδώ ε, αντιβαίνει στις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι ε, μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ε, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες στις οποίες πρέπει να συμμετέχουν και οι πολίτες και αυτό δεν έγινε. Πολλά στοιχεία αυτής της αναφοράς αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, τη δημοσία υγεία, τα κριτήρια βιώσιμης κινητικότητας, πολλές αιτίες για να διατηρηθεί ανοιχτή αυτή η αναφορά και πολλές αιτίες για να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη στιγμή που θα έρθει η γραπτή απάντηση. Πείτε μας κάτι πιο ρητό, κάτι πιο συγκεκριμένο, κάτι πιο αποτελεσματικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Σλάιν. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ ήθελα να ευχαριστήσω τους αναφέροντες. Ήταν πολύ δομημένη, πολύ ακριβή αυτή η αναφορά. Στην Πολόνια το συζητούν αυτό εδώ και καιρό. Πολύ συχνά μας λένε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Η μηδενική επιλογή δεν εξετάστηκε καν. Αντιθέτω, είμαι πεπισμένη ότι πάντα υπάρχει εναλλακτική, πάντα πρέπει να υπάρχει. Ε, έστω και η πολιτική βούληση να υπήρχε, αλλά από ό,τι φαίνεται αυτή η λύπη Δεν υπάρχει πολιτική βούληση να ακολουθεί κάποια άλλη οδό. Εγώ θέλω να στηρίξω απόλυτα τι επιτροπέ που παρακολουθούν το θέμα επιτόπου και που θέτουν εύλογα ερωτήματα. Συμφωνώ με τον συναδέλφο Αφρόντε. Η απάντηση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων δεν μπορεί να είναι τόσο επιφανειακή. Δεν μπορούμε ε, να ανοίπτουμε τα σχέδια μας όπως ο Πιλάτος ε, ελπίζοντας οι αρχές των κρατών μελών να επιβάλλουν ε, τήρηση ευρωπαϊκών οδηγιών ειδικότερα όταν μιλάμε για θέματα διαφάνειας, συμμετοχής όλα αυτά δεν μπορούν να παραμένουν στα χαρτιά μόνο ειδικότερα σε εποχές όπου αντιμετωπίζουμε μια κρίση εμπιστοσύνης δυσπιστίας μάλλον προς τα ευρωπαϊκά όργανα πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να δώσουμε μια σωστή απάντηση άμεσα ε, για αυτό το έργο το οποίο ανησυχεί τους πολίτες από πολλές απόψεις. Δεν φαίνεται να επιλύεται το ζήτημα της ε, υπερβολικής κίνησης στην περιφερειακή οδό ε, και της σχετικής ρήπανσης. Φαίνεται ότι περισσότερο έχει γίνει μια προπαγάνδα, μια διαφήμιση αποφάσεων που έχουν ήδη ληφθεί. Ε, και που θέλουμε να γίνουν δεκτέ απλά από του πολίτε, να τι επιβάλλουμε στου πολίτε, κάτι που δεν μπορούν να δεχτούν οι πολίτε. Όταν είναι τόσο δεινέ οι επιπτώσει στην υγεία του και στο περιβάλλον, όπω ε, ακούσαμε μάλιστα, πρόκειται για μία από τι πιο μολυσμένε περιοχέ τη Ιταλία. Αυτό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, όπου στην Ιταλία όπου το μοντέλο προωθείται είναι ένα απερχαιωμένο. Ε, εξακολουθούν να επενδύουν στο τσιμέντο, στις, ε, στους περιττούς αυτοκινητοδρόμους και στην υποβάθμιση του εδάφους. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν θαραλέες επιλογές που να οδηγήσουν σε μια μεγάλη αλλαγή προς ένα πιο βιώσιμο μοντέλο. Κλείνω ε, παραλαμβάνοντας την υποστήριξή μου στηρίζοντας την έκκληση της συναδέλφου Εύη να παραμείνει ανοιχτή αναφορά και το πρόβλημα να εξεταστεί προσεκτικά από την Επιτροπή αυτή του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει επίση και οι Ιταλικές αρχές να συλλέξουν πιο πολλά και ακριβή δεδομένα ε, περί τη ρήπανση ε, στην, ε, στο περιφερειακό της Μπολόνια διότι με τα στοιχεία που υπάρχουν σήμερα δεν μπορούν να ληφθούν αποφάσεις σωστές για το μέλλον εμάς των κατοίκων της Μπολόνια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Ιέκα. Να ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα εστιαστώ σε δύο βασικά θέματα. Αφενός ε, έχουμε ένα ευρωπαϊκό ε, πλαίσιο που προτείνει περιβαλλοντικά αναπτυξιακά μοντέλα, μοντέλα επενδύσεων ε, με γνώμονα την προστασία της υγείας των πολιτών αλλά και του περιβάλλοντος προσεγγίζουμε μια στρατηγική ε, όπου το 2050 στόχος είναι να έχουν μειωθεί οι εκπομπές ε, και ε, να βελτιώσουμε τα εδάφη. Αντιθέτως, τοπικά παρατηρούμε ότι αυτά τα σχέδια για το μέλλον αποτελούν το αντικείμενο απόλυτης παράβλεψης. Σήμερα η υποβάθμιση του εδάφους είναι κάτι που δεν συζητείται ειδικότερα ε, και παρότι ζητείται μια καλύτερη στρατηγική για την χρήση του, ε, κινούμαστε αντιθέτως προς μια τσιμεντοποίηση, όλο και μεγαλύτερη. Έχουμε έργα τα οποία καταστρέφουν το περιβάλλον στην Ιταλία. Ε, το περιβάλλον, τη φύση που αποτελεί ανθρώπινη κληρονομιά για ολόκληρη την ανθρωπότητα και ούτε δίνουμε αρκετή προσοχή στο θέμα της προστασίας των Υγεία της υγείας των πολιτών. Πολλοί κάτοικοι της Μπολόνια ζουν μόνιμα σε μια ατμόσφαιρα ανθυγιεινή. Υποχρεούνται να αναπνέουν μολυσμένο αέρα. Είναι ένα σοβαρό το πρόβλημα το οποίο πρέπει να επιληθεί. Οι στρατηγικές με τις οποίες θα πρέπει να αξιοποιήσουμε όλους τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας ε, βελτιώνοντας για παράδειγμα το σιδηροδρομικό δίκτυο, την ε, κοινή χρήση αυτοκινήτων, ε, συγκοινωνίες που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όλα αυτά τα προγράμματα πρέπει να επιτέλους να εφαρμοστούν. Να υπογραμμίσω ότι έχουμε σχεδόν 650 εκατομμύρια ευρώ τα οποία έχουν επενδυθεί σε αυτό το έργο. Και θέλω να πω απλά τι θα μπορούσε να γίνει αν χρησιμοποιούσαμε όλους αυτούς τους πόρους και υλοποιούσαμε ε, ε, βιώσιμες μεταφορές που να σέβονται όχι μόνο το περιβάλλον και τα εδάφια αλλά και την υγεία κυρίως των πολιτών. Το αίτημα λοιπόν της συναδέλφου Εύη και το δικό μου αίτημα είναι να διατηρηθεί ανοιχτή αυτή η αναφορά αλλά και η Ιταλική κυβέρνηση για πρώτη φορά ενδεχομένως σε αυτό το τομέα επιτέλους να ξυπνήσει να ξυπνήσει από το λίθαργο, να ξεκινήσει επιτέλους ε, ε, έργα με γνώμονα την υγεία των πολιτών. Αυτά τα καταραμένα έργα που υποβαθμίζουν ε, το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών θα πρέπει να σταματήσουν να είναι τόσο πολύ αριθμό σε τόσο πολλά εργοτάξια. Είναι τεράστια η καταστροφή που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια από τέτοια έργα η Μπολόνια αξίζει κάτι καλύτερο. Βιώσιμες μεταφορές, ε, βιώσιμες συγκοινωνίες, μια ένα στρατηγικό όραμα επενδυτικό που να καθησυχάζει τις ανησυχίες των πολιτών με τρόπο αηφόρο. Τα 657 εκατομμύρια που θα χρησιμοποιηθούν για το έργο αυτό θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή εκατοντάδων βιώσιμων έργων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση αυτή η Ιταλο-Ιταλική και τώρα περνάμε στην Ισπανο-Ισπανική. Κύριε Κάμπρας. Ευχαριστώ. Δεν συμφωνώ απόλυτα με τους συναδέρφους οι οποίοι μίλησαν. Συμφωνώ απόλυτα με τους συναδέλφους που μίλησαν. Ε, να βάλουμε έτσι ένα δρόμο στη μέση της Μπολόνια αν κατάλαβα καλά, μιλήσετε για 65 εκατομμύρια, όχι 650 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Όχι. 65 εκατομμύρια οχήματα το χρόνο. Τεράστια ποσότητα. Τεράστιος αριθμός. Και το να κάνουμε πιο φαρδί τον αυτοκινητόδρομο, κατανόητο τελείως είναι ένα έργο το οποίο είναι επιβλαβές για τους πολίτες. Οι συνάδελφοι αναφέρθηκαν στην υγεία. Είναι κάτι σημαντικό φυσικά. Αλλά αυτό που εμένα μου κάνει τεράστια έκπληξη είναι η Κομισιόν που λέει ότι, ότι μεταξύ άλλων πρέπει να λάβουμε υπόψη τον κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Μεταξύ άλλων. Μα τι λέτε. Αυτό έπρεπε να είναι το πρώτο που θα μας απασχολεί. Η ανθρώπινη υγεία είναι μια πρωταρχική αξία, δεν είναι απλά μια αξία μεταξύ των υπολείπων. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι το ζήτημα του περιβάλλοντος δεν είναι κάτι μόνο εξωτερικό. Το ζήτημα του περιβάλλοντος ξεκινάει από το σπίτι μας, από το δρόμο μας, από τη δουλειά μας. Εξού και συμφωνώ απόλυτα. Η αναφορά πρέπει να παραμείνει ανοιχτή. Ευχαριστώ πολύ. Okay. Uh, thank you to all of... Ε, σας ευχαριστώ όλους όσοι συμμετείχατε σε αυτή την συζήτηση και τώρα επανέρχομαι κύριε Τασινάρη σε εσά. Δύο λεπτά έχετε ακόμα στη διάθεσή σας εφόσον το επιθυμείτε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εμένα μου κάνει έκπληξη τα όσα είπε η Κομισιόν. Φαίνεται ότι προερχόνται μόνο από μια οπτική γωνία. Δεν φαίνεται να αξιολόγησαν τα πράγματα που απασχολούν εμά. Όσον αφορά τη συμμετοχή, η συμμετοχή είναι κάτι που πρέπει να γίνεται στην αρχή τη διαδικασία, όπω λέει η συνθήκη του όρχου. Δεν μπορείτε να έρχεστε και να, να, να μας λέτε ότι η διαβούλευση για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι η μόνη ε, στιγμή ε, συμμετοχής των πολιτών που μπορεί να μας παραχωρηθεί. Εμείς πρέπει να συμμετέχουμε κατά την ε, λήψη της απόφασης της στρατηγικής απόφασης για το περιβάλλον. Αυτό το έργο, σε αντίθεση με όλα τα σχέδια εδαφικού προγραμματισμού των μεταφορών στην Εμίλια Ρωμάνια, στην αστική περιοχή της Μπολόνια, έρχεται σε αντίθεση με τα πάντα. Η συμμετοχή έπρεπε να γίνει τη στιγμή που θα αποφασιζόταν τι θα γίνει, όχι αφού έχει αποφασιστεί τι θα γίνει. Και η ρήπανση ε, λένε ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Πηγαίνετε να δείτε ε, τι έχουν μετρήσει τα κέντρα φέτος. Είναι δραματικά τα αποτελέσματα, δραματικές οι μετρήσεις. Δεν μπορείτε να μου λέτε ότι βελτιώνεται η ποιότητα του αέρα. Έχουμε μετρήσει έως και πενταπλάσια από τα ανεκτά επίπεδα. Και αυτή τη στιγμή μέσα σε έξι μήνες 20 φορές έχουμε υπερβεί τα όρια. Άμα ε, ε, μιλάτε και μιλάτε για βελτίωση του αέρα στην Πολόνια. Ο αέρας στην Πολόνια είναι φρικτός. Οι, οι, οι υγειονομικές επιπτώσεις δεν έχουν μελετηθεί. Το, τις έχει ζητήσει ε, η περιφέρεια της Εμίλα Ρωμάνια και το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν τις παραχώρησε. Οπότε παρακαλώ να ενημερώνεστε πλήρως για τα όσα συμβαίνουν σχετικά με αυτό το έργο, διότι αυτό που συμβαίνει είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν μπορείτε να μιλάτε για εκτιμήσεις ε, υγειονομικών επιπτώσεων, διότι η περιφερειακή οδός στην Πολόνια δεν περιλαμβάνει ε, σημεία ελέγχου των ρήπων. Ε, κάτι που ζητάνε οι πολίτες εδώ και χρόνια. Οπότε σας παρακαλώ, ε, πραγματικά ως ευρωπαϊκά όργανα εμβαθύνετε λίγο την επιχειρηματολογία, λάβετε πληροφορίες από όλου, όχι μόνο από την Ατοστράντε Περλιτάλια και από την Ιταλική κυβέρνηση, δείτε πιο αναλυτικά θέματα που αναφέρονται και στην αναφορά αυτή. Δείτε και την έκθεση ε, που έχουμε προσαρτήσει στην αναφορά, ε, έκθεση που αφορά το Πασάντε την Πολόνια. Ελπίζω να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά, διότι εμείς ε, βασιζόμαστε στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε και εγώ, εύχομαι να παραμείνει η αναφορά ανοιχτή και ευχαριστώ όλους τους προαναλύσαντες. Τα όσα είπαν ε, κινούνται προς σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να υπογραμμίσουμε πόσο παράλογο είναι αυτό το έργο το οποίο προβλέπει διαπλάτηση ενός αυτοκινητοδρόμου ο οποίος περνά ε, ε, σε απόσταση 10 μέτρων από μέρη όπου κατοικούν άνθρωποι. Ευχαριστώ. 10 μέτρα από τα σπίτια των ανθρώπων και ξέρουμε την πολιτιστική κληρονομιά και τη σημασία που έχει η πόλη της Μπολόνια. Οπότε και αυτό πρέπει να το λάβουμε πολύ υπόψη. Δεν πρόκειται μόνο για την περιφέρεια, για την πόλη, για την Ιταλία την ίδια. Είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα για όλους μας. Γιατί είναι ένα κομμάτι της Ευρώπης που ανήκει σε όλους. Ωραία. Θα μείνει ανοιχτή λοιπόν και θα περιμένουμε τη γραπτή απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο μεταξύ θα στείλουμε επιστολή στις Εθνικές και Περιφερειακές Αρχές της Ιταλίας όπου θα επιμένουμε ότι παρακολουθούμε το ζήτημα. Αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε. Έτσι, ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστούμε που ταξιδέψατε μέχρι τις Βρυξέλλες για να μας τα πείτε όλα αυτά. Να επιστρέψετε με ασφάλεια πίσω στην Πολώνια. Καλό ταξίδι. Επόμενη αναφορά. Δεν έχουμε εδώ την αναφέρουσα, δεν εμφανίστηκε ακόμα. Ίσως να είναι στο δρόμο, δεν ξέρω. Μπορούμε να περάσουμε έτσι στο επόμενο θέμα, που είναι η γνωμοδότηση σχετικά με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα άτομα με αναπηρίες. Και είναι πολύ απλό, διότι εγώ είμαι η συγκήτρια για τη γνωμοδότηση αυτή. Οπότε σας ε, παρακαλώ να με παρακολουθήσετε λίγο. Λοιπόν, ξέρετε ότι όταν ασχολούμαστε με αυτήν την ε, στρατηγική, η αρμόδια επί επιτροπή είναι η Επιτροπή Επασχόλησης. Η δικιά μας όμως η συμβολή είναι να βασίσουμε τη δικιά μας γνωμοδότηση στις αναφορές, στις σχετικές που έχουμε πάρει. Αυτό δίνει μια προστιθέμενη αξία στην τελική έκθεση γιατί κατοπτρίζει και τις απόψεις των πολιτών. Οι αναφορές λοιπόν που έχουμε πάρει μέχρι τώρα υπογραμμίζουν την ανάγκη να υπάρξει μια οριζόντια προσέγγιση για άτομα με αναπηρίες και την πρόσβασή τους σε διάφορα αγαθά. Οπότε, εμείς βασιζόμαστε στο άρθρο 9 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία και επιμένουμε ότι πρέπει να εφαρμοστεί συνολικά έτσι ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δημόσια αγαθά και υπηρεσίες όπως εσείς και εγώ. Στη γνωμοδότησή μου λοιπόν τονίζω δύο ζητήματα πάνω στα οποίο έχουμε δουλέψει πολύ στην Επιτροπή μας. Το ένα είναι η εφαρμογή της συνθήκης του Μαρακές και το δεύτερο είναι το δικαίωμα όλων να μπορούν να ζήσουν ως ανεξάρτητα άτομα στο σπίτι τους. Αυτό σημαίνει ότι οι χώρες μέλη πρέπει να τηρήσουν την αρχή και τη διαδικασία της αποειδηματοποίησης και να διευκολύνουν αυτή τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στις κοινοτικέ υπηρεσίες, όπως ε, το είδαμε με την περίπτωση της Σλοβακίας πέρυσι. Προσβλέπω στην συμβολή όλους, όλων σας και ελπίζω ότι στο τέλος θα εγκρίνουμε τη γνωμοδότηση αυτή, η οποία πιστεύω θα βοηθήσει στην βελτίωση και στον εμπλουτισμό της τελικής έκθεσης. Τώρα, βάσει της Επιτροπής Απασχόλησης το κείμενο της γνωμοδότησης είναι μόνο στα αγγλικά και ό,τι τροπολογίες έχετε πρέπει να υποβληθούν μόνο στα αγγλικά. Λυπάμαι γι' αυτό, αλλά δεν εξαρτάται από μένα. Δεν είχα τη δυνατότητα να το αλλάξω. Έχει να κάνει με την Επιτροπή Επασχόλησης και το δικό του χρονοδιάγραμμα. Είναι πάντως σημαντικό να στείλουμε τη γνωμοδότησή μας Λοιπόν, προθεσμία για υποβολή τροπολογιών είναι αύριο Τετάρτη. Στις 12... Όχι, στις 3. 3 διορθώνει η Πρόεδρος. 5 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Θα πάρετε βέβαια και πρόσκληση, αλλά να το σημειώσετε ότι η πρώτη συνάντηση σκιωδών προβλέπεται ήδη για την 5η Σεπτεμβρίου. Αυτά. Σχόλια. Παρακαλώ κύριε Τερικάμπρες. Ευχαριστώ. Η προθεσμία είναι τρει αύριο, έτσι, σωστά, κατάλαβα. Ωραία, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόταση γνωμοδότησης όσον αφορά την εφαρμογή της στρατηγικής για τα άτομα με αναπηρίες. Η έκθεση πρόοδου αντικατοπτρίζει τις προκλήσεις οι οποίες παραμένουν τα πλαίσια της στρατηγικής αυτής της Ευρωπαϊκής. Η Επιτροπή μας έχει ήδη παραλάβει διάφορες αναφορές που έχουν να κάνουν ε, με την ε, δυνατότητα πρόσβασης και θα ήθελα να προσθεθεί και αυτό, να τονιστεί και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, η ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρίες και ο ρόλος της υπηρεσίας αυτής, του οργανισμού αυτού, προκειμένου να διευκολύνει την εφαρμογή της σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Γι' αυτό θα υποβάλω φιλικές τροπολογίες από αυτού. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Πολύ ωραία. Καλά ακούγεται. Ωραία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Η κυρία Κρούνα. Ή όχι. Όχι. Όχι. Λάθος. Λάθος έκανα το όνομα. Η κυρία Πορέρο, σωστά. Ωραία, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Πλαθέτια Πορέρο ονομάζομαι. Ευχαριστώ την Επιτροπή σας. για την γνωμοδότηση αυτή που ετοίμασε. Πράγματι αναφέρονται ήδη πολλά σημαντικά στοιχεία στην γνωμοδότηση αυτή που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή της σύμβασης του ΟΗΕ και την έκθεση πρόοδου βάσει των αναφορών που έχετε ήδη παραλάβει. Τώρα, όπως αναφέρεται και στην έκθεση πρόοδου, θέλω να σας πω ότι τα δύο ζητήματα στα οποία αναφερθήκατε, η προσβασιμότητα πρώτα απ' όλα, είναι όντω κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουμε αφιερώσει ιδιαίτερη προσοχή. Θέλω να επενθυμίσω μάλιστα την πρόταση για την ευρωπαϊκή πράξη δυνατότητας πρόσβασης, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη κάνει πολλά ώστε να δει το θέμα αυτό της δυνατότητας πρόσβασης συνολικά και με τρόπο που να επηρεάζει θετικά και να βοηθάει τα άτομα με αναπηρίες. Τώρα για το δεύτερο θέμα της ανεξάρτητης ζωής των ατόμων αυτών, προβλέπουμε στους κανονισμούς των διορθωτικών ταμείων κάποια ενίσχυση στην διαδικασία αυτή μετάβασης από την ιδρυματική ζωή σε ανεξάρτητη ζωή με βοήθεια από την κοινότητα. Είμαστε στη διάθεσή σας γιατί ό,τι άλλες διευκρινήσεις χρειάζεστε και σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, εμείς σας ευχαριστούμε. Υπάρχει απόλυτη συνοχή από ό,τι βλέπω μεταξύ των θεσμικών οργάνων σε αυτή την περίπτωση. Πολύ καλό. Ωραία. Αμφανίστηκε άλλη μια συνάδελφος, η κυρία Μπεσέρα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ ε, για τη γνωμοδότησή σας, που είναι πολύ επίκαιρη. Αντικατοπτρίζει όντως πολύ καλά τη συνοχή που υπάρχει μεταξύ των θεσμικών ε, οργάνων. Η Επιτροπή Αναφορών έχει μεγάλη σημασία ακριβώς γιατί επεξεργάζεται τις διάφορες αναφορές που μας φτάνουν στα πλαίσια της σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία. Ό,τι δουλειά έχουμε κάνει μέχρι τώρα, τονίζει ακόμα περισσότερο την ανάγκη οι δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών να παραμένουν ζωντανές και να τους δίνεται προβολή γιατί αντικατοπτρίζει τις απόψεις και τους προβληματισμούς των πολιτών. Το θέμα αυτό για την πρόσβαση ατόμων με προβλήματα όρασης, για παράδειγμα, σε όλα τα δημοσιευμένα έργα, είναι κάτι θετικό και βοηθάει να τηρήσουμε την αρχή της μη διάκρισης. Χρειάζεται ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για να ευνοηθεί η κοινωνική ένταξη των ατόμων αυτών. Από πλευρά των φιλελεύθερων προτείνουμε να προσθέσουμε ότι πρέπει γρήγορα να ακυρωθεί η συνθήκη του Μαρουέκος που σχετίζεται βέβαια με τη σύμβαση του ΟΗΕ και με την διακήρυξη την οικουμενική για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Το τελευταίο για την συνθήκη του Μαρακές υπάρχει ήδη στη γνωμοδότησή μου. Οπότε όντω υπάρχει μεγάλη συνοχή και μεταξύ μας και πρέπει να είμαστε περήφανοι που για χρόνια εδώ στην Επιτροπή μας τονίζουμε την ανάγκη κύριο της συνθήκης του Μαρακές. Λοιπόν τώρα, τι θα προσπαθήσω να κάνω με τη γνωμοδότηση. Θα προσπαθήσω να υπογραμμίσω τον ε, ρόλο προστασίας που έχει η Επιτροπή μας Και θα αναφερθώ επίσης και στο μεγάλο αριθμό αναφορών που μας στάνουν κάθε χρόνο και που αναφέρονται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν Ευρωπαίοι πολίτες παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε τα δύο κεντρικά ζητήματα είναι η δυνατότητα πρόσβασης, βέβαια, και το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα. Εννοείται που χαίρομαι πάρα πολύ που ε, επιτέλους αναβαθμίσαμε λίγο αυτό το θέμα. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Αύριο μέχρι τις 3 έχετε περιθώριο για την υποβολή τροπολογιών. Και η πρώτη συνάντηση σκιωδών εισηγητών θα είναι 5 Σεπτεμβρίου, μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Και η ψηφοφορία θα γίνει εδώ, στην Επιτροπή μας, στις 7 Σεπτεμβρίου. και 19 Οκτωβρίου θα ψηφίσει η Επιτροπή Απασχόλησης. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα λοιπόν που έχουμε μπροστά μας. Και λυπούμε που πρέπει να πω τώρα ότι αναφέρουν που έχει να κάνει με την κατασκευή δεξαμενής ρύθμισης για τον ποταμό Σεβέζο δεν είναι εδώ. Οπότε θα αναβάλουμε αυτό το σημείο. Για κάποια άλλη στιγμή, ίσως για το απόγευμα, δεν ξέρω. Τώρα τίποτα άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε γιατί δεν είναι εδώ. Α, μια στιγμή. Ωραία. Μου ήρθαν κάτι νέα για την αναφέρουσα. Είναι στο δρόμο από το αεροδρόμιο Σαρλερουά. Δεν πρόκειται να δω σε λίγα λεπτά όμως, οπότε αυτήν την αναφορά θα την εξετάσουμε πρώτη στις 3. Να είσαστε εδώ στις 3 και θα αρχίσουμε με αυτή την αναφορά. Σας ευχαριστώ πολύ.